Πού πάει πού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 Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitamme. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε τις εργασίες της Υποπιτροπής αυτής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Arvoisat läsnäolijat, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλώς ήρθατε όλοι σε αυτήν την συνεδρίαση της Υποεπιτροπής μας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σήμερα το κύριο θέμα μας θα είναι ακρόαση που έχουμε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Θέλω εδώ να κηρύσω την έναρξη των εργασιών μας, ε, ζητώντας σας καταρχήν εγκρίνετε το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε? Ωραία. Δεύτερο σημείο. Γνωρίζουμε ποιο θα είναι ο τέταρτος αντιπρόεδρος της υποβιτροπίσ μας. Οι σοσιαλδημοκράτες όρισαν τον κύριο Γιάννου Τσέμπκεν. Υποθέτω ότι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Οπότε, εφόσον συμφωνείτε, σας ζητάω να εγκρίνουμε την εκλογή του ως τέταρτος αντιπρόεδρος της υποπιτροπής μας. Καλώς, ωραία. Καλώς ήρθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μάλλον αγαπητέ συνάδελφε, ελάτε εδώ μαζί μας, στο Προεδρείο και ερχόμαστε στο τρίτο σημείο πρακτικά της προηγούμενης συνεδριάσεως της 31ης Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου 2009. Εγκρίνονται τα πρακτικά? Ωραία, εγκρίνονται. Και τώρα περνάμε στο σημείο 4. Κάποιες ανακοινώσεις έχω να σας κάνω από πλευράς της Προεδρίας σχετικά με το τι έγινε εκ μέρους της υποπιτροπής μας τις εβδομάδες που πέρασαν. Πρώτα απ' όλα, για τον πρόεδρο Σαντρίκενεν και εγώ ίδια συντάξαμε επιστολή σχετικά με το Ιράκ, Κάνε Ραφ, ο υπουργό Εξωτερικών της ε, στον Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδική Προεδρίας. Του ζητάμε να οργανώσει τα πράγματα έτσι ώστε να μπορέσει μια ομάδα παρατηρητών του ΟΗΕ να πάει στο Καραντάσρα η κυρία Αντρίκενεν και εγώ ίδια πριν από μερικές εβδομάδες στείλαμε έτοιμα, ζητούσαμε δηλαδή από την Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ να δράσει. Αυτά λοιπόν που κάνουμε εδώ στην Υποπιτροπή μας είναι απόλυτα στην γραμμή που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του του Μαΐου για την ανθρωπιστική κατάσταση των ε, κρατουμένων ε, στο στρατόπεδο ΑΣΡΑΦ. Θέλουμε πληροφορίες περισσότερες για την κατάσταση εκεί. Από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα για όσους βρίσκονται εκεί. Γι' αυτό και ζητήσαμε από τη Σουηδία να δράσει και να φροντίσει να λυθεί το πρόβλημα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Στη συνέχεια, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπήρξε ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκε. 17 Σεπτεμβρίου, από την άλλη μεριά, εγκρίναμε ψήφισμα για την περίπτωση για εκβέκνη που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν. Πρόκειται για έναν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, ξέραμε ότι ο κύριος Τσόφτ δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από μια δίκαια δίκη. Η δίκη αυτή που έγινε εναντίον του που είχε να κάνει με το θάνατο ενός πεζού σε κάποιο τροχαίο ε, μας δείχνει ότι υπάρχουν ε, πολιτικές πτυχές εκεί. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε από τις αρχές του Καζακστάν να ε, μελετήσουν ανοιχτά το θέμα αυτό, να ερευνήσουν τι ακριβώς έγινε και να δημοσιοποιήσουν τις λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, γιατί το Καζακστάν είναι η χώρα που αναλαμβάνει την Προεδρία του ΟΑΣΕ το 2010. Και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υπενθυμίσουμε στο Καζακστάν τις υποχρεώσεις που έχει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι ε, το Συμβούλιο Σύνδεσης με το Καζακστάν ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεδριάσει μέσα Νοεμβρίου. Τότε θα ξέρουμε φαντάζομαι περισσότερα. Κάτι άλλο τώρα από την επικαιρότητα, ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε στο Στρασβούργο και είχε να κάνει με τον Μοχάβετ Αλχασάν, Σύριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τις Συριακές Αρχές την άμεσα απελευθέρωση του ανθρώπου αυτού που είναι εμπειρογνώμων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της οργάνωσης Σουασί ε, που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυλακίστηκε στις 28 Ιουλίου, είναι πρόεδρος αυτής της οργάνωσης και κατηγορήθηκε ότι υπονομεύει την ασφάλεια του Συριακού κράτους. Ε, στη συνέχεια ότι διέδωσε ψευδείς ειδήσει. Διάφορα, διάφορες κατηγορίες, οι οποίες όμως δεν ακούστηκαν ξεκάθαρα προς τα γιατί όλα έγιναν και κλεισμένο των θυρών. Ένα άλλο θέμα επικαιρότητα, πάλι ένα άλλο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει να κάνει με τη δολοφονία άλλου που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, δίχως άλλο. Τι άλλο. Α, ναι. Συναντήθηκα με πολλούς εκπροσώπους από το Συμβούλιο της Ευρώπης τη βδομάδα που ήμασταν στο Στρασβούργο. Και είμαι πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να διατηρήσουν στενές σχέσεις μεταξύ τους. Και να τις κάνουμε μάλιστα ακόμα πιο στενές. Και αυτό για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα μεταξύ μας. Μπορούμε ίσως να συζητήσουμε μαζί κάποιες δράσεις. Για παράδειγμα, 20 χρόνια του βραβείου Σαχάροφ ή 20 χρόνια από τότε που πέθανε ο ίδιος ο Σαχάροφ. Ίσως θα μπορούσαμε από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης να οργανώσουμε κάτι για αυτή την επέτειο. Κάτι άλλο. 22 Οκτωβρίου έχουμε μία επιπλέον συνεδρίαση έκτακτη της υποπιτροπής μας. Και αυτό για να συνδεθούμε με τον Τούμα Σαμπανό που είναι ε, αρμόδιος ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι μια έκτακτη συνεδρίαση, σημειώστε την παρακαλώ. Θα μας δοθεί έτσι ευκαιρία να συζητήσουμε και πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο Σαχάροφ. Κάτι άλλο. Συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Τρεβ Στίβενσεν, ο οποίο είναι υπεύθυνο για την ε, καταπολέμηση των βασανιστήριων, πάντα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για το θέμα αυτό λοιπόν, που έχει να κάνει με την αναξιοπρεπή μεταχείριση ε, και τα βασανιστήρια. τα μέλη, προβουλευτές δηλαδή και το Προεδρείο της Υποβιτροπής μας ε, έχουν πάρει πρόσκληση για μια διάσκεψη που γίνεται στις 6 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια. Στη συνεδρίαση αυτή θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι από την Νομική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ελπίζω, υποθέτω, ότι σας ενδιαφέρει το θέμα. Θα μας δοθεί έτσι ευκαιρία να έχουμε πιο στενή συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την καταπολέμηση των βασανιστήριων. Τέλος, θέλω να σας πω ότι η πρόθεσή μας είναι να οργανώσουμε συνάντηση ή συναντήσεις στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Ντίκ Μάρτιν. Ο Ντίκ Μάρτιν δεν δουλεύει πια για τη ε, μεταφορά ε, εξοδικαστικά κατηγορούμενων, αλλά Δεδομένου ότι η προσωρινή επιτροπή που είχε φτιαχτεί και είχε ασχοληθεί με αυτές τις πτήσεις της CIA, νομίζω ότι θα μας ενδιαφέρε να δούμε λίγο και μαζί του τι έγινε από τους ηθήνοντες. Υπάρχουν πολλά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Πάρα πολλοί ζητούν να συναντηθούν μαζί μας. Πάντως, σε αυτό που θέλω να επιμείνω είναι ότι έγιναν συζητήσεις με την ομάδα για τη Βερμανία δηλαδή. Έχω έρθει σε επαφή με διάφορες οργανώσεις και προσπαθώ να δω πώς θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τις εκλογές που θα γίνουν στη Μιαμάρα σε λίγο, που οργανώνει η Χούντα Υπάρχει πολύ χαμηλή αξιοπιστία βέβαια όσον αφορά αυτές τις εκλογές, οπότε πρέπει να δούμε τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε εν ώψη των εκλογών αυτών. Ξέρω ότι σας είπα πολλά. Όμως έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε και να περάσουμε στο πέμπτο μας σημείο που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Και εδώ δεν χρειάζεται να σας πω ότι η Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια έχει ιδιαίτερα δραστηριοποιηθεί και παρακολουθεί την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Αυτά τα θέματα εδώ στην Υποπιτροπή μας συζητιούνται πάρα πολύ συχνά. Θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Το καλοκαίρι είχαμε δολοφονίες υποστηρικτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άντρε Γκουαγκίν, Νατάλια Στεμίροβα, η κυρία Σαντολάγεβα, Άλικ Τσελάγεβιτς. Αλίκ Μπάιλο, Αναστάσια Βαμπαμπούροβα, Πάρα πολλά ονόματα, τα οποία ε, βλέπουμε ότι χάνονται σιγά σιγά. Οι άνθρωποι αυτοί χάνονται και στο Βόρειο Κάφκασο. Η κατάσταση είναι καταστροφική. Σε αυτήν λοιπόν εδώ την ακρόαση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να επικεντρωθούμε στην κατάσταση στον, στον Βόρειο Κάφκασο. Σε ένα πρώτο στάδιο λοιπόν αυτό που θα ήθελα είναι να ζητήσω από, τρεις, από τους τρεις ομιλητές που έχουμε να μας μιλήσουν 10 λεπτά περίπου ο καθένας. Πρέπει να επενθυμίσω ότι οι βουλευτές μας θέλουν πάρα πολύ να ακολουθήσει και συζήτηση. Γι' αυτό σας παρακαλώ και τους τρεις να περιοριστείτε στο χρόνο που σας δίνουμε, ώστε μετά να μας δοθεί ευκαιρία να έχουμε πραγματικά συζήτηση μεταξύ μας, γιατί είναι που μας ενδιαφέρει όλους. Έχουμε και μια σύνδεση Skype με τον Στάνισλαβ Δημητρίευσκη. που είναι διευθυντής ε, αρχιστάκτης ε, της εφημερίδας Πραβοτσάστικα πίσεις έχει γράψει κάτι για τα εγκλήματα στη Τζεζενία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έκθεση. Στα αγγλικά υπομορφή βιβλίου, δεν ξέρω πού ακριβώς. Πάντως οι ευρωβουλευτές μπορούν να το έχουν στη διάθεσή τους. Έχει μοιραστεί. Βέβαια χρειάστηκε δυστυχώς να χρησιμοποιήσουμε το Skype για να έρθουμε σε επαφή με τον Στάνισλαφ Δημητριεύσκη γιατί του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Δημητριεύσκη. Καλώς ήρθατε στην υποπιτροπή μας αυτή. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε διερμηνία. Σας το λέω αυτό να το ξέρετε από τα ρωσικά. Τι κάνετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση αυτή της Υποπιτροπής μας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Δημητριευσκή. Θα ήθελα 10 ε, λεπτά τώρα, λέει η Πρόεδρος, να σας δώσω για να μας παρουσιάσετε ε, την κατάσταση, δηλαδή να μας πείτε τι είναι αυτό που είναι σημαντικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Το γεγονός ότι έχετε προσκληθεί σε αυτή την συνεδρίαση δείχνει ότι περιμένουμε από εσά να μας ενημερώσετε. Έχουμε στη διάθεσή μας έγγραφα που έχετε ετοιμάσει εσείς και οι δύο άλλοι προσκεκλημένοι μας. Και τα έχουμε. Λοιπόν, 10 λεπτά σας δίνω το λόγο και μετά ελπίζω να είσαστε στη διάθεσή μας να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου λοιπόν καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο σε αυτή τη σύνδεση. Όσον αφορά την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά στη Ρωσία και ειδικότερα στο Βόρειο Κάφκασο, πρέπει να σας πω ότι οι διεθνείς οργανώσεις μιλούν για ευθύνη του κράτους. Αλλά η ευθύνη του κράτους είναι στην πραγματικότητα ευθύνη συλλογική. Θα έπρεπε να μιλήσουμε μάλλον για συλλογική ανευθυνότητα. Και για να υποστηρίξω τη θέση μου αυτή μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ήδη εγκρίνει πολλά ψηφίσματα για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την Τσετσενία, όπου εμπλέκεται η Ρωσία όσον αφορά την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως, το υπεύθυνο για αυτά κράτος τι κάνει, πληρώνει τα πρόστιμα που επιβάλλει το δικαστήριο, χωρίς όμως να καθορίζεται κάποιο ω υπεύθυνο και χωρίς να διώκεται κανένας υπεύθυνο. Η ατιμορρησία επικρατεί. Τα εγκλήματα λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό και στη Ρωσία μιλάμε για την ε, πληρωμή των χρημάτων αυτών από πλευράς ε, της Ρωσίας σαν να πρόκειται για φόρο που επιβάλλει η Ευρώπη όταν πρόκειται για κλιματικές ενέργειες. Η διεθνής κοινότητα λοιπόν πρέπει να καταδείξει τους υπευθύνου ως άτομα και όχι ως κράτη. Ακόμα και αν αυτό είναι δύσκολο, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάτε. Η οργάνωσή μας ε, ολοκλήρωσε μία μελέτη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Βόρειο Κάφκασο. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε εκεί διάφορα κείμενα δικαίου, την ομολογία επίσης διεθνών δικαστηρίων, σε περιπτώσεις όπως ήταν η Ιουγκοσλαβία ή η Ρουάντα. Καταλήξαμε στα εξή συμπεράσματα αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη μας. Τα εγκλήματα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τους πολέμους στην Τσετσενία δεν ήταν απλώς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν ήταν απλώς παραβιάσεις της ρωσικής νομοθεσίας. Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα εγκλήματα αυτά έγιναν από τους δύο κύριους εμπλεκόμενους στον πόλεμο, υπεύθυνοι από πλευράς της Τσετσενίας, που οι περισσότεροι έχουν πεθάνει, ή ε, τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις ή έχουν εξαφανιστεί, ενώ υπεύθυνοι από πλευράς της Ρωσίας παραμένουν σε ατιμορρησία. Οι ρωσικές αρχές ποτέ δεν οργάνωσαν καμία έρευνα για τα εγκλήματα αυτά ούτε καν για μασικές δολοφονίες ε, πληθυσμού στη Τσετσενία. Οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν πάντα να προβούν σε τέτοιου είδους έρευνες και μελέτες και μάλιστα οργάνωσαν και συγκεκριμένες ενέργειες για να στηρίξουν τη στρατιωτική τους δράση εκεί. Στείλανε διάφορα τάγματα θανάτου σε πολλές ε, περιοχές όπου βρίσκονται άοπλοι. Ρωσικές αρχές λοιπόν, όπως σας είπα, αρνήθηκαν πάντα να ερευνήσουν τέτοια θέματα και πάντα αρνήθηκαν τις ευθύνες τους όσον αφορά τους ε, στρατιώτες που πάνε εκεί. Είναι λιγάκι σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα που είναι υπέρ πάσης υποψίας πάντα. Οι ρωσικές αρχές λοιπόν δεν θέλουν να συνεργάζονται όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας αναγκάζει να αναφερόμαστε εδώ στο θέμα της ε, οικουμενικής ευθύνης και αρμοδιότητας. Καταλαβαίνετε ότι οι ευθύνες βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο ε, στρατιωτικών εντολών. Έχουμε και μάλιστα πολλές αποδείξεις από αυτού και έχουμε πολλές αποδείξεις για το ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα πολιτισμένων λαών παραβιάζονται. Η υπεύθυνη είναι πολύ βέβαια. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τον Βλαντίμιρ Πούτιν που είναι σήμερα πρωθυπουργό και για τον Ζορ Κατηρόφ, το θέατρο της Τσετσενίας και τον Σαμανόφ του κατά τσεφ και για πολλούς πολλούς άλλους που είναι λίγο πολύ γνωστοί. Όλοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα κατά ε, του πληθυσμού και προσπάθησαν να μας ε, πείσουν ότι ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που έκαναν. Αν μη τι άλλο είναι ηθικά υπεύθυνοι για τις εντολές που έδωσαν. γιατί είναι συνένοχοι, συμμετείχαν σε εγκληματικές δράσεις όλη αυτή την περίοδο. Το 2003 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με το ψήφισμα 1326 είπε ότι εφόσον το κλίμα αυτό ατιμορρησίας εξακολουθήσει στην Τσετσενία, τότε η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο να βρει τους υπεύθυνους οργανώνοντας ένα ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα στην Τσετσενία. Δυστυχώς μετά το ψήφισμα αυτό τίποτα δεν έγινε. Έχει περάσει τόσο καιρό, αλλά ούτε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ούτε και τα άλλα όργανα του Συμβουλίου της ε, Ευρώπης έκαναν κάτι για να θέσουν σε εφαρμογή αυτό το ψήφισμα. Έτσι όπως έχει η κατάσταση λοιπόν σήμερα, οι Ρώσοι ηγέτες, το σημερινό κλίμα διεθνών σχέσεων είναι τέτοια που η δημιουργία ενός τέτοιου δικαστηρίου είναι κάτι το αδύνατο. Όμως τα πράγματα αλλάζουν, εξελίσσονται. Ε, Μιλόσεβιτς, Καράζεβιτς, ε, Πινοσέτ ε, κλπ. είναι περιπτώσεις που μας κάνουν να ελπίσουμε ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές και να είναι εφικτή λύση αυτού του ειδικού δικαστηρίου. Ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει την πρωτοβουλία που δεν πήραν οι υπεύθυνοι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει μια ερευνητική επιτροπή για την κατάσταση στην Τσετσενία. Φυσικά τέτοιου είδου επιτροπές ξέρω ε, μελετάνε το πράγμα και υιοθετούν εκθέσεις οι οποίες όμως στη συνέχεια ποτέ δεν τίθεται σε εφαρμογή. Όμως ξέρω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά να βρεθούν ε, τα στοιχεία, οι αποδείξεις και έτσι να δημιουργηθεί αν μη τι άλλο μια βάση δεδομένων για την κατάσταση στη Τσετσενία. Θα μπορούσατε να εμπνευστείτε από την Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ε, το ψήφισμα 780 όσον αφορά τα εγκλήματα που έλαβαν χώρα στην τέο Γιουγκοσλαβία. Θα μπορούσατε να εμπνευστείτε από αυτό. Βέβαια δεν λέω ότι θα υπάρξει συνεργασία με τις ρωσικέ αρχές. Θα είναι δύσκολο να στείλετε αποστολές παρατήρησης επιτόπου σύντομα. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αν μη τι άλλο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις που θα μπορούσαν εκείνες να οργανώσουν έρευνες επιτόπου στο Βόρειο Κάφκασο. Σύμφωνα με τις ε, προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν και στην προηγούμενη επιτροπή σας και τα θύματα και οι ε, διάφορες μαρτυρίες που θα μπορέσετε να συλλέξετε θα βοηθήσουν. Πολλοί έφυγαν από την Τσετσενία εδώ και 10 χρόνια και έχουν εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Η Επιτροπή δεν πρέπει να βάλει προθεσμίες. Είναι μια δουλειά που, όπως έλεγα και πριν, θα κρατήσει πολύ. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, είναι απαραίτητο η δουλειά αυτή να γίνει με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ισχύει μια πολύ προθυμένη νομοθεσία όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, προσπάθησα να σας παρουσιάσω σύντομα την υπόθεσή μας, αλλά είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στανισλάβ, για την παρέμβασή σου. Μας επιτρέπει να σκεφτούμε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα ότι δηλαδή σε όλο τον κόσμο και στο Βόρειο Κάυκασο οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να καταγραφούν με έναν τρόπο ώστε οι ένοχοι να προσέλθουν στη δικαιοσύνη. Στις Βρυξέλλες ελπίζουμε η υγεία σας να παραμείνει καλή εκεί που είστε. Γιατί έχουμε δει ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου απλή. Καλό θα είναι να συναντηθούμε όσο πιο σύντομα γίνεται είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Σαζούργο ή και στο Ελσίνκι και το, τα έγγραφα που έχετε συγκεντρώσει είναι ιδιαίτερως χρήσιμα θα ήθελα να παραμείνετε παρόν στη συζήτηση, να πάρετε μέρος και στο υπόλοιπο τμήμα. Τώρα θα δώσω το λόγο σε Σεργέη Κοβαλιόφ, ο οποίος ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την εποχή του Μπόρις Γέλτσιν, ο οποίος εκρατήθη κατά επανάληψη Βλέπω ότι ο κύριος Κοβαλιόφ μου γνέφει. Εγώ καλωσορίζω τον κύριο Κοβαλιόφ εδώ και θα ήθελα να μας μιλήσει. Έχουμε όμως το όνομα της Καρίνα Μοσκολέγκο. Θα θέλαμε να είναι παρούσα, αλλά και αυτή είναι στη Μόσχα δεν ήρθε. Παρακαλώ λοιπόν τον Σαργέη Κοβαλιόφ να αυτοπαρασιαστεί. Υπήρξατε πολιτικό κρατούμενο στη Σοβιετική περίοδο ω υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότερο από όλου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσφατα έγραψα μία επιστολή στον πρόεδρο Μετβέντεφ και το ρώτησα γιατί η πολιτική βία στρέφεται μόνο κατά της αντιπολίτευσης, αυτών που είναι κατά της κυβέρνησης. Γιατί συμβαίνει αυτό. συμφωνείτε με τους ληστές ή κάνετε αυτό που ο Στάλιν είπε για τους ε, κοινωνικούς φίλους ή για τους εγκληματίες αδελφικούς φίλους. Φυσικά στο ερώτημά μου απάντηση δεν πήρα. Μετά όμως ήρθε ένας αστυνομικός στο σπίτι μου με μια επιστολή και σε αμηχανία του είπε ότι οι ανώτεροι του τον επιφόρτησαν να απαντήσει στην επιστολή μου αλλά δεν ήξερε πώς να απαντήσει στην επιστολή μου. Τα συζητήσαμε λοιπόν και αποφασίσαμε και ότι και οι δυο μας βρισκόμαστε σε αμήχανη δύσκολη θέση για κάποιον άγνωστο λόγο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου συμφώνησα με ένα αστυνομικό. Φυσικά οι ερωτήσεις μου πιθανώς δεν ήταν προσβλητικές. Πάντως δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Οι γραφειοκράτες της κυβέρνησης προσπάθησαν τάχα να απαντήσουν στις ερωτήσεις μου Ίσως θα ήθελα να μου πούνε ξέρουμε πότε πρέπει να σκοτώσουμε κάποιον. Οι πολιτικές εκτελέσεις των αντιφρονούντων της αντιπολίτευσης είναι πια ένα μαζικό φαινόμενο. Υπάρχει μια μακρά λίστα ονομάτων. Βίκτωρ Παπκόφ, Ζούρα Μπετιέφα. Ιβλόιφ, Ναταλία а Зарема Садулаева, Умар Джабраилов. Это последние жертвы. Αυτά είναι τα τελευταία θύματα, τα πιο πρόσφατα θύματα που δολοφονήθηκαν πρόσφατα. Και αυτό δείχνει ποια είναι η πολιτική της ρωσικής κυβέρνησης. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα ονόματα στη λίστα. που ζουν πολύ δύσκολες καταστάσεις στο Βόρειο Κάφκασο Αγκαλιάς. τα же Άννα Πολιτκόφσκα και Νατάλια Стемирова отнюдь не узкокавказского звучания персоны – ε, ε, ε, Όλα τα ονόματα αυτά είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τον Κάφκασο. Λιτβινιένκα, Στανισλάβ Μαρκέλοφ. Вот и ένας μακρύς κατάλογος που δεν είναι όμως πλήρης και ποτέ δεν θα ολοκληρωθεί για τον απλούστατο λόγο ότι Ποτέ δεν θα ξέρουμε πώς να ταξινομήσουμε, πού να ταξινομήσουμε αυτούς που τους έχουν απαγάγει, που εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν πίσω ίχνο ζωής ή τον οποίον το, ε, ε, το πτώμα βρέθηκε σε μαζικούς τάφους ή που το του κόμπε και το κεφάλι από έκρηξη χειροβομβίδας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι πολιτική βία και πολιτικών δολοφονιών. Και εδώ μιλάω για ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στο Βόρειο Κάφκασο και σε μεγάλες πόλεις. Τι μπορούμε όμως να πούμε για τα θύματα που δολοφονήθηκαν σε άλλα τμήματα της χώρας, άτομα τα οποία δηλητηριάστηκαν με αέριο. που υπήρξαν θύματα εκρήξεων στη διάρκεια μαχών. Μιλάμε για εκατοντάδες θύματα. Σας θυμίζω ότι τα θύματα των εξήκρεσεων, των εκρήξεων σε διαμερίσματα στη Μόσχα είναι και αυτά θύματα. Δεν ξέρουμε τι θύματα είναι. Δεν ξέρουμε αν το σκότωσαν τρομοκράτες από τη Βόρεια Κάυκασο ή αν τους σκότωσαν ε, Ρώσοι σπίτσνας ή ειδικέ υπηρεσίες. Δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε. Μιλάμε όμως για πολλές εκατοντάδες θυμάτων και σας θυμίζω τα, ε, τα τάγματα θανάτου στην Τσετσενία, τα εκτελεστικά αποσπάσματα. Και έχουμε εδώ αποδείξεις ότι πρόκειται για κρατική τρομοκρατία. Φυσικά θα ήταν φυσιολογικό να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με το πώς η κυβέρνηση ασκεί το νόμο στη χώρα αυτό που καλεί σύνταγμα που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ένα ενεργό σύνταγμα αλλά στην πραγματικότητα ένα σύνταγμα που δεν εφαρμόζεται. Δεν έχουμε ελεύθερες εκλογές Έχουμε λογοκρισία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει καταμερισμός στις εξουσίες. Και θα πρέπει να διερωτηθούμε σε τι βαθμό αυτή η χειραγώγηση όσον αφορά το, το δίκαιο και το Σύνταγμα σχετίζεται με τα θύματα της πολιτικής τρομοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς κρατούμενους και πάλι μεταξύ των οποίων και ο παδί του Λεμόνοφ ξέχασα το όνομα ξέχασα το όνομα του κομματός είναι πάρα πολύ ενεργοί στη δράση τους και σίγουρα δεν τους αξίζει, δεν τους αξίζει να κρατούνται στη φυλακή επί έτη, να τιμωρούνται από την κυβέρνηση με διοικητικά μέτρα. Έπειτα οι επιστήμονες μας, πολλοί επιστήμονες στη Ρωσία, όπως γινόταν με την κλασική σοβιετική παράδοση, φυλακίζονται για κατασκοπία. Γι' αυτό σας θέτω αυτό το ερώτημα. Σε τι βαθμό αυτό σχετίζεται με τις πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία. Σε τι βαθμό οι πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία σχετίζονται με την Ευρώπη. Εμείς, εμείς εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην καρδιά της Ευρώπης. Και η Ευρώπη θα ήθελα να είναι μία Ευρώπη, ενωμένη Ευρώπη. Και μάλιστα το θέλει αυτό αποφασιστικά. σε ερωτώ λοιπόν. Αυτή η κρίση που εμείς θεωρούμε πολιτική, νομική και ηθική κρίση σε τι βαθμό επηρεάζει αυτή η κρίση στην Ευρώπη. Εγώ απαντώ, επηρεάζει πάρα πολύ. Ο Στάβνη Σταυρντιμητριεύσκη και εγώ μιλήσαμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Αναφερόμαστε μάλλον σε αυτά τα όργανα και σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι στο ψήφισμά του για την κρατική τρομοκρατία στην Τσετσενία το κοινοβουλευτικό αυτό όργανο πρότεινε ορισμένε αποφάσει οι οποίε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Παραδείγματο χάρη, μία απόφαση λέει να υπάρχει μία διαδικασία προκειμένου να στερηθεί το καθεστώς μέλους της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Επειδή όμως οι αποφάσεις στο Συμβούλιο παίρνονται με ομοφωνία, υπήρξε δυσκολία. Το ψήφισμα έχει και ένα άλλο σημείο, το οποίο έλεγε ότι τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έπρεπε να στραφούν κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο στο Στρασβούργο. Ποια χώρα το έκανε αυτό, ποια χώρα έκανε αυτή την προσφυγή, καμία. Ρώτησα τους πολλούς φίλους στην κοινοβουλευτική συνέλευση γιατί και μου είπανε «Μα καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε, ε, αισθανόμαστε άσχημα να διαμαρτυρόμαστε γιατί η Ρωσία». Είναι σαν να αρχίζουν να ξαναμαλώνουν οι παλιές σλάβικες φυλές μεταξύ τους. αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό αυτής της συνολικής κρίσης που επαναλαμβάνω δεν είναι η οικονομική κρίση. Έχω ακόμα 60 δευτερόλεπτα νομίζω στη διάθεσή μου. Συνεχίζω λοιπόν. Επαναλαμβάνω, δεν είναι οικονομική κρίση, είναι μια ιστορική, ηθική και αν μου επιτρέψετε θα μπορούσα να προσθέσω και νομική κρίση. Γι' αυτό οφείλω να δηλώσω ότι εκτιμώ πολύ τα δημοσιεύματα του Αξένσο Πανιτσεύσκη και Δημητριεύσκη είναι πάρα πολύ χρήσιμη η δουλειά τους, πάρα πολύ λεπτομερής και χρήσιμη. Θα ήθελα ταυτόχρονα να προσθέσω ότι η προσωπική ευθύνη δεν είναι ίδια με την ευθύνη του κράτους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι οι διεθνείς αποφάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα μας λένε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γνωρίζουν σύνορα. είναι θέμα υπερσυνοριακό. Αυτό είχα, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ την προσοχή σας ότι δεν πρέπει να έχω μόνο θρησκευτικά τελετουργικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ομιλία. Προφανώ και το ζήτημα εδώ δεν είναι απλώ μια οικονομική κρίση και οι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία δεν θα πρέπει να γίνονται αντιληπτέ ω ε, μια κρίση οικονομική φυσή. Εμεί θα θέλαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα για την κρίση του Βορειού Κάφκασου. Γι' αυτό είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε μαζί μα, τον κύριο Χάσκη, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση στην Οικουσετία Και βέβαια σε τέτοιου είδου αυταρχικά καθεστώτα ακριβώ η αντιπολίτευση δεν έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή τη. Και ο και ήταν ε, και εκείνο στην Κουσατία. ήταν αρμόδιος σε ζητήματα σε σχέση με το διαδίκτυο και είχε δολοφονηθεί τέσσερις ημέρες μετά από την παρουσία του εδώ στις ε, Βρυξέλλες. Δεν θέλαμε εδώ να τον τιμήσουμε για μία ακόμα φορά. Κύριε Χάσμα, θα θέλαμε να ακούσουμε από εσά πώ έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Οικουσιατία κατά τη δική σα άποψη. Έχετε το λόγο, κύριε Κασπίεφ. meeting. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πρέπει να σας πω ότι όλοι προσπαθούν να συμμετάσχουν. έτσι ώστε να προληφθούν περαιτέρω πολιτικές ε, δολοφονίες. Δηλαδή μιλάμε, συζητάμε και δύο εβδομάδες αργότερα δολοφονούνται και άλλοι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω πως αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει εάν ε, δεν κάνουμε κάτι από την ολόκληρου του κόσμου. Ε, και εδώ ε, στην τελευταία περίπτωση είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα γιατί γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο υπέτειος, ποιος είναι ο αυτούργος. Στις προηγούμενες περιπτώσεις δεν γνωρίζαμε, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Ο Πρόεδρος ε, κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών και ο Υπουργός Εσωτερικών ε, ε, μπήκε στο αυτοκίνητό του και προβολήθηκε στο κεφάλι και μετά πετάχθηκε στον δρόμο. Έχουμε μετά μια συνάντηση, συζητούμε, δύο εβδομάδες αργότερα δολοφονούνται και άλλοι. Τώρα, τι συμβαίνει στην Ιγκουσετία. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω το τι συμβαίνει. Είναι απερίγραπτο. Θα πρέπει να μεταβείτε εκεί και να δείτε με τα μάτια σας το τι συμβαίνει. Κατά έξι χρόνια κατά το οποίο ο κύριος Ζάσκοφ ήταν ο πρόεδρος, είχαμε ομάδες θανάτου οι οποίες μένονταν στους δρόμους. Οι αρχές δεν έκαναν τίποτα για αυτές τις ομάδες και κανένας δεν μιλούσε για αυτές. 2.000 άνθρωποι ηλικίας ε, μικρότερες από 20 ετών δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας του, ενώ πολλοί άνθρωποι αγνοούνται, εξαφανίστηκαν, ενώ ο κύριος Ζάζεκ ε, συναντιόταν με τον κύριο Πούτιν και του έλεγε ότι εγώ κατασκευάζω βιομηχανίες, κατασκευάζω κατοικίες και ούτω καθεξής. 70 νέε επιχειρήσει ακούσαμε ότι δημιουργήθηκαν. Τι, τι έγινε εκεί, κάποιο θαύμα, τίποτα δεν έγινε. Ε, Όμω τέτοιε αναφορέ έκανε ο πρόεδρο των ε, Πούτιν, αλλά κανένα δεν είδε τελικά αυτέ τι επιχειρήσει στην Εκουσιατία. Μάγκο ο δημοσιογράφος δηλαδή ο οποίος δολοφονήθηκε, είχε ε, αναφερθεί σε αυτό ε, και έχει αυτογραφίσει επανειλημμένα γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα ε, φοβόμαστε. Θα συνεχίσουμε δηλαδή να ενημερώνουμε τη κοινή γνώμη σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Προφανώ δεν υπάρχουν ανεξάρτητε εφημερίδε ή περιοδικά, αλλά έχουμε μια πολύ καλή ιστοσελίδα και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για το πώ έχουν τα πράγματα στην Οικουσετία. Θα πρέπει μια ανεξάρτητη επιτροπή να οργανωθεί για να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση έρχονται αντιπροσωπείε στην οικουσετία, συναντιόνται με τον πρόεδρο, πίνουν μαζί του τσάι και στη συνέχεια γίνουν στι πατρίδε του, χωρί να συμβαίνει τίποτα. Ε, οι αντιπροσωπείε αυτέ, οι επισκέπτε θα πρέπει να συναντηθούν με εμά, να, να δουν κανονικού άνθρωπου, να μιλήσουν με οικογένειε των οποίων μέλη έχουν εξαφανιστεί, να μιλήσουν με, άνθρωπα, ε, με ανθρώπους συγγνώμη, οι οποίοι βασανίστηκαν εγώ πρόσφατα επισκέφτηκα το πλοίο που είναι ένα μικρό χωριό, και ε, μίλησα με μια οικογένεια, της οποίας ε, ο γιος ε, απήχθη. Και η αστυνομία είπε στους γονείς ότι θα, τον, θα μετέβαινε σε ένα αστυνομικό κέντρο στην Ικουσετία. Αυτό δεν συνέβη. το μεταφέρανε στην Τσετσενία όπου και βασανίστηκε για 24 ώρες δεν μπορεί πλέον κανείς να δει αυτό το αγόρι. Είναι απίστευτο. Τον βασάνισαν ε, με ηλεκτροσόκ, ε, τον έκοψαν ε, με μαχαίρια. Δηλαδή είναι απερίγραπτο, ήταν, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί σε τι κατάσταση ήταν. Δεν μπορεί κανεί να φανταστεί δηλαδή τι είδου βασανιστήρια υπέστη. Ο καμεραμάν ο οποίο βρισκόταν εκεί άρχισε να κλαίει. Και δεν ξέρουμε γιατί, γιατί τον βασάνισαν. Ε, λένε σχετικά, του είπαν πε μα το όνομα ενός ε, τρομοκράτη. Ε, μα έλεγε ποιον, οποιονδήποτε. Υπήρχαν κάποιε ρωσικέ αρχέ και του είπαν πε μα ένα όνομα, ποιο θα μπορούσε να είναι τρομοκράτης, ένας γείτονα, ένας φίλος, οποιοδήποτε. είναι πραγματικά απίστευτο. Πριν από κάποιο καιρό ήμουν στο Παρίσι και διαπίστωσα ότι υπάρχουν 8.000 πρόσφυγες εκεί. Από την Ιγκουσετία. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν, να φύγουν από την Ιγκουσετία. Και γι' αυτό σας είμαι ευγνώμων που με καλέσατε σήμερα εδώ για να μου δώσετε τη δυνατότητα να εκφραστώ την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ στις Βρυξέλλες σήμερα. Και πραγματικά σας απευθύνω έκκληση να μην σταματήσετε. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Χάσβιε, για αυτά που μας είπατε που πραγματικά σοκάρουν. Εγώ να κάνω μια πρόταση. Δεδομένου ότι θα συζητήσουμε τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα ήθελα να στήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Προεδρία του Συμβουλίου, τη Σουηδία, να εκφραστούν επ' αυτού. Η κατάσταση έχει ως εξή. Η διάσκεψη Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία θα λάβει χώρα 18 ε, και 19 Νοεμβρίου. Και ως ήθιστε, θα γίνουν και συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 4 με 5 Νοεμβρίου. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να έχουμε στοιχεία, δεδομένα, για να τα χρησιμοποιήσουμε στη διάσκεψη. Καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει να έχουμε διαβουλεύσεις, συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πηγαίνουμε στη διάσκεψη κορυφής μάδια τα χέρια, σαν να μην τρέχει τίποτα. Γι' αυτό θέλω να στήσω από τον Γιάννη Μουτλάντερ που είναι πρέσβης για τα ανθρώπινα δικαιώματα από πλευράς της Προεδρίας. Κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε εδώ. Ξέρω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη Σουηδία είναι προτεραιότητα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παίρνω το λόγο στην υποπιτροπή σας. Θα ήθελα να αναγνωρίσω ότι οι μαρτυρίες που ακούσαμε είναι πάρα πολύ σοβαρές του κύριου Δημητριεύσκη, του κύριου Χασπιεύ και του κύριου Κοβάλιεφ. Θα ήθελα συγχρόνως, κυρία Πρόεδρε, να τονίσω εδώ ότι η Προεδρία του Συμβουλίου δίνει ιδιαίτερη προσοχή και χτυπάει το κουδούνι του συναγερμού κάθε φορά που ακούει περιπτώσεις όπου πλήττονται τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στην ε, Ρωσία όσο και στον Βόρειο Κάφκασο. Στο Βόρειο Κάφκασο αναμφίβολα έχει αυξηθεί η βία τα, τους τελευταίους μήνες. Ίσως να έχετε διαπιστώσει μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει δημόσια τις πρόσφατες βιότητες και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία. Η Σουδική Προεδρία λοιπόν έκανε ανακοίνωση καταδικάζοντας την ε, δολοφονία της κυρίας Εστιμόρεβα μετά την απαγωγή της και τον Αύγουστο υπήρξε και δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δολοφονίες της κυρίας Αντουλάγεβα και του συζύγου της Τζαμπράιλερ ζητήσαμε έρευνα σε βάθος των δολοφονιών αυτών από τις ρωσικές αρχές. Επιπλέον, το Σεπτέμβριο εκφράσαμε βαθιά ανησυχία στο μόνιμο συμβούλιο του ΟΑΣΕ για δολοφονία του κύριου Μπλουμάλη Καχμεντήλοφ στο Πακιστάν. Στο Πακιστάν. Και αυτό προκειμένου να συνεισφέρουμε στο τέλος της περίοδου ατιμορρησίας, στην οποία τόσο καλά αναφέρθηκε ο κύριος Δημήτριευσκη και όπως και εκείνος έζησε και εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος αυτό. Όμως να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρησιμοποιήσει και έναν άλλο δρόμο για να χειριστεί τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτές είναι οι διαβουλεύσεις που έχουμε με την Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα που λαμβάνουν χώρα μία φορά ανά κάθε Προεδρία. Την τελευταία φορά ήταν τον Μάιο στις Βρυξέλλες και ο επόμενος γύρο θα λάβει χώρα αρχές Νοεμβρίου στη Στοκόλμη. Οι συναντήσεις αυτές, των συναντήσεων αυτών προηγούνται συναντήσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εμείς, η Σουηδική Προεδρία, θα συνεχίσουμε αυτή την πρακτική, αυτή την παράδοση. Έχει Ήδη γίνει μια τέτοια συνάντηση και θα υπάρξει και άλλη μια ακριβώς πριν τις διαβουλεύσεις με την Ρωσία. Οι συζητήσεις μέχρι τώρα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, είχαν σαν θέμα τη λειτουργία της κοινωνίας, η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία συνεταιρίζεστε, η ελευθερία όσον αφορά ε, όπως είπαμε, την έκφραση, η καταπολέμηση των διακρίσεων, ε, των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. κλπ. Πολύ σημαντικό επίσης είναι εδώ να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να βάζει θέμα και όσον αφορά ατομικέ περιπτώσεις με τη Ρωσία. Και έχουμε πάρει κάποιες απαντήσεις για την τύχη ανθρώπων που είχαμε συμπεριλάβει στον καταλογό μας. Για τη Στοκόλμη συζητάμε την ημερήσια διάταξη ακόμα με τη Ρωσία. Δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμα έξι εβδομάδες μπροστά μας. Θα ήθελα όμως να σας πω ήδη από τώρα, νομίζω ότι μπορώ, ότι προτείναμε ένα ειδικό θέμα για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφκασο. Όπως επίσης και θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. Συνεπώς, κυρία Πρόεδρε, θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και θα συνεχίσουμε επίσης να αναφέρουμε και ατομικές περιπτώσεις και να ζητάμε εξηγήσει για αυτές από τις ρωσικές αρχές. Είμαστε ανοιχτοί επίσης ε, στα briefing αυτά ε, μαζί σας, με τα μέλη της Υποπιτροπής δηλαδή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς μπορούμε να σας στείλουμε καταλόγους με υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων η υγεία ή η ζωή έχει τεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους. Έτσι μπορείτε πιο αποτελεσματικά να συζητάτε για αυτά τα θέματα με τις ρωσικές αρχές. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπόθεση αυτή. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κύριος Τίμανς, είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αποδώσω φοροτιμής στους Ρώσους φιλοξενούμενους μας, πολλοί από τους οποίους τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ και χρόνια από στενή συνεργασία στα πλαίσια της προετοιμασίας για τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαίωματα, Πολλούς από αυτούς επίσης τους ξέρουμε και στα πλαίσια υποστήριξης προγραμμάτων που χρηματοδοτούμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να επαναλάβω αυτό που εξήγησε η Πρόεδρος όσον αφορά τη διαδικασία και φυσικά η Κομισιόν συνεργάζεται με τη διαδικασία αυτή. Η κατάσταση στη Ρωσία είναι αρκετά σοβαρή και θα έπρεπε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Από τη μια μεριά, οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας πρέπει να επικυρωθεί και από το Ευρωκοινοβούλιο και σε αυτό το πλαίσιο θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα παίξουν μείζωνα ρόλο ιδιαίτερα όσον αφορά να υπάρξει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία στην αρχή αυτής της συμφωνίας. Δεν ασχοληθήκαμε ακόμα με αυτή την πτυχή στις διαπραγματεύσεις. Θα φτάσουμε όμως και σε αυτό. Και αυτό θα είναι, παραπάνω ένα μείζον θέμα στις ε, σοβαρές συζητήσεις, στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία σε, στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο της Ένωσης, δηλαδή η προσεχή διάσκεψη κορυφής το Δεκέμβριο και στις τακτικές ε, διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις ρωσικές αρχές και να επιμείνουμε, να εμείνουμε, να τηρήσει τις υποχρεώσεις της η Ρωσία με βάση τη συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης και με βάση τις ε, συμφωνίες των Ηνωμένων Εθνών. Μερικές φορές παραξενευόμαστε, είμαστε από τη μια μεριά έχουμε δημόσιε δηλώσει και που τι κάνει και ο πρόεδρος Μετβέντεφ ο ίδιος κατά του νομικού μηδενισμού όπως τον χαρακτήρισε που βασιλεύει στη Ρωσία και από αυτό συμπεραίνουμε ότι, ότι λαμβάνονται μέτρα από τη διοίκηση. Από την άλλη μεριά τα γεγονότα με τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τα φασανιστήρια όπως ακούσαμε πριν, είναι μια πραγματικότητα. Κάτι δεν πάει καλά. Είτε υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, είτε υπάρχει αβελτηρία όσον αφορά στον ε, μηχανισμό της δημόσιας ασφάλειας. Πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση στο Βόρειο Κάυκασο, στην Τσετσενία, την Ιγκουσετία και στον Ταγκεστάν καθέα αυτή έχει μια δική της δυναμική που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την ιστορία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αφενός να το δούμε συγκεκριμένο το θέμα αυτό και με ρωσικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με την αντιπροσωπεία μας στη Μόσχα και με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει τρόπος να βοηθήσουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί που διατρέχουν κίνδυνο συγκεκριμένα. Τι δυνατότητα υπάρχει να τους δοθούν ε, προσωρινά βίζες εύκολα το συζητάμε και μεταξύ μας και με τις κυβερνητικές οργανώσεις, τι δυνατότητα έχουμε να αυξήσουμε κατά κάποιο τρόπο μέσα προσωπικής προστασίας. με ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις που προστατεύουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε κονδύλια που θα μπορούσαμε να θέσουμε στη διάθεσή τους. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Διερευνούμε όλα αυτά που σας ανάφερα, επειδή η κατάσταση χειροτερεύει. Από την άλλη μεριά τώρα, δεν θα ήμασταν ε, έντιμοι με τους εαυτούς μας σχετικά με το τι πίεση μπορεί να ασκήσει η Ένωση στη Ρωσία. Αν πούμε ότι είναι απεριόριστη. Είναι περιορισμένη. Μπορεί να θέσουμε ορισμένα θέματα. Και η πρόεδρος το είπε. Πόσο ευθέως θα πρέπει να καταδικάσουμε τις δολοφονίες και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Αλλά τελικά την ευθύνη την έχει η ρωσική κυβέρνηση και οι ρωσικές αρχές αυτές πρέπει να πάρουν μέτρα. Πολιτικά, αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να υπενθυμίσουμε τις ευθύνες που έχει η ρωσική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, σε πολιτικό επίπεδο κυρίως. Δεν μπορούμε όμως να παρεύουμε και να δράσουμε εμείς αντί για τη ρωσική, τις ρωσικές αρχές. Πώς μπορούμε λοιπόν τώρα να βοηθούσουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κινδυνεύουν. Το πιο συγκεκριμένο που μπορούμε να κάνουμε πέρα από τα πολιτικά μηνύματα που πρέπει να περνάμε σε όλα τα επίπεδα προς τις ρωσικές αρχές είναι αυτό που σας ανάφερα πριν. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τίμανς. Φυσικά και εσείς και ο κύριος Νόλαντερ, ο πρεσβευτής, ξέρουμε ότι δουλεύετε συνεχώς. Πάντως η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία δεν έδωσε αποτελέσματα. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Είπατε ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει στο ύψιστο δυνατό επίπεδο. Αυτό όμως δεν συγκεκριμενοποιείται, ακόμα και αν εσείς ή εγώ ή κάποιος άλλος το θέλουμε. Πρέπει πραγματικά να υπάρξει κάποια επίπτωση. Σας αναγνωρίζω το ότι αναγνωρίζετε την υπόθεση υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντω, η Ένωση πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο. Καλό ήταν τότε να φέρατε κάτι συγκεκριμένα, συγκεκριμένα μέτρα. Και τώρα Ας δώσουμε τη δυνατότητα στους συναδέλφους, βουλευτές, να μιλήσουν. Και οι προσκεκλημένοι μας, που είναι και στην πρώτη σειρά καθισμένη, η κυρία Βιντάλ, ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, η κυρία Τσελούσεβα, που συνεργάστηκε με τον Στανιστάβ Δημητριεύσκη, με όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία ακούσαμε γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα στη Ρωσία έχουμε τον Αντρέι Νεκρασόφ στην πρώτη σειρά σκηνοθέτη ο οποίος έκανε ένα φιλμ που το είδαμε χθε για τον πόλεμο Ρωσίας-Γεωργίας και έχουμε και τους συναδέλφους. Καταρχήν δίνω το λόγο στα μέλη της αντιπροσωπείας για τη Ρωσία. Ποιος θέλει το λόγο. Καλό θα είναι τα μέλη της αντιπροσωπείας για τη Ρωσία παρόντες. Ο πρώτος δυστυχώς ε, είχε ένα κόλλημα, δεν είναι παρόν. Ο κύριος Μπέρμαν λοιπόν πρώτος. Θα ήθελα να μιλήσω ρώσικα, αλλά νομίζω πως έχει πολύ, περάσει πολύ στήρος αυτό το Δεν τα έχω μιλήσει λοιπόν για πολύ πολύ καιρό. Είναι μια πολύ όμορφη γλώσσα, αλλά δεν μπορώ να τη μιλήσω πολύ καλά. Ως ανταποκριτής λοιπόν στη Μόσχα για το Ολλανδικό ραδιόφωνο, είχαμε την, ε, την νέα αντίληψη ότι σταδιακά με την ελεύθερη αγορά η ανάγκη για κράτος δικαίου θα ανέκυπτε. από την ίδια την ανάγκη δηλαδή του να ότι σε σεβασμού τα συμβόλαια και γενικά να ότι σε σεβασμού οι νόμοι. Αυτός ε, όμως αυτή η αισιόδοξη ε, αντίληψη μετά από όλη την θριαμβευτική κατάρρευση του τείχους και ούτω καθεξής ε, ε, κατέρευσε και αυτή. Δηλαδή ουσιαστικά δεν βρισκόμαστε σε καμία περίπτωση σε κράτος δικαίου. Σε κράτος ατιμορρησίας βρισκόμαστε. Εγώ είχα τη δυνατότητα να συναντηθώ με την δημοσιογράφη κυρία Άννα για πολλές φορές και ήμουν στους σοσιαλιστικής πολιτική ομάδα είχα αφήσει και λουλούδια στο, στον τάφο της ε, ε, με μεγάλη μου λύπη ε, και όταν είχα ρωτήσει τον συντάκτη της Νοβαγιακαζέτα Καζέτα τι πρέπει να γίνει βέβαια αυτή είναι και η αιώνια πολιτική φράση πάντως μου είχε απαντήσει ότι μην μας στείλετε χρήματα θα θεωρηθούμε ως συνεργάτες σας και αυτό μπορεί να, με τη σειρά του να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για να μας τι να εκδίδουμε την εφημερίδα μας. Αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε πάρα πολύ προγράμματα με Ρώσους φοιτητές και Ρώσους δημοσιογράφους ώστε να δουν το τι σημαίνει ανοιχτή δημοκρατία αφού τους στερείται το δικαίωμα να ζουν μέσα σε μια τέτοια ανοιχτή δημοκρατία. Εάν λοιπόν ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι, και αυτό βέβαια φαίνεται λίγο αστείο στα κοινικά μάτια του Κρεμλίνου, είναι να έχουμε τέτοιου είδους προγράμματα ανταλλαγής και να ανοίξουμε τα σύνορά μας για τους Ρώσους φοιτητέ, επιστήμονες, δημοσιογράφους, ώστε να μπορέσουν να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε στην δημιουργία δημοκρατικής συνείδησης. Κύριε θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για κάτι τέτοιο. Είναι μια πολύ μικρή, αν θέλετε, περιορισμένη πρόταση σε σύγκριση με τα όσα πραγματικά χρειάζεται η Ρωσία. Ε, και κάτι ακόμα θα ήθελα να προσθέσω. Δεν με την απεσιοδοξία σας ως προς την ηθική κρίση και τη δικαστική κρίση στον κόσμο γενικά. Εάν έχουμε ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο, τότε ε, μπορώ να πω πως αν σημειώνεται κάπου πρόοδος είναι ακριβώς στον τομέα της δικαιοσύνης. Η, αυτή καθεαυτή η ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σημαίνει ότι οι αρχηγοί κρατών δεν μπορούν πλέον να θεωρούν ότι θα βρίσκονται σε καθεστώς ατιμορρησίας ή τουλάχιστον ε, η ύπαρξη του δικαστηρίου καταδεικνύει ότι δεν θα πρέπει να ζουν σε ατιμορρυσία. Αλλά προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι ερχόμενος από τη Μόσχα είσαστε έτσι λίγο απεσιόδοξος θλιμμένο σε σχέση με αυτό. Όμω ε, μια πρόοδο σαν αυτή νομίζω πως υπάρχει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπέρμαν. Ε, θα δώσω αργότερα στον κύριο Κοβάλεφ. Ε, ζητώ συγγνώμη κύριε Κοβάλεφ. Θα ακούσουμε κάποια ερωτήματα και συνέχεια θα δώσουμε το λόγο σε εσά για να απαντήσετε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ραλόχπηδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ακούσαμε πολύ γλαφύρες περιγραφές της κατάστασης όταν ακούσαμε δηλαδή ότι υπάρχουν ομάδες θανάτου ε, και καθώς Ρωσία ε, όπως είπε και ο κύριος Κοβάλεφ αποτελεί περιφερειακή δυναμική για μας για την Ευρώπη θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο γενικά, όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της ενέργειας και ούτω καθεξής και όχι μόνο να περιοριζόμαστε σε δηλώσεις σε καλές ε, Ο πρόσωπος της Οικουσιασίας μας είπε ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που θέλουν να φύγουν από εκεί ε, και εκεί θα πρέπει να επιδείξει την διάθεση, τη βούληση η Ευρώπη να αποδεχτεί άτομα από αυτές τις περιοχές, αλλά έχουμε ε, βιώσει την εμπειρία ε, πολλές φορές να απελάβνονται άτομα τα οποία μεταβαίνουν στην Ευρώπη. Το βιώσαμε και με τη Ζεσενία αυτό. Ε, δηλαδή υπενθυμίζω την υποχρέωση που έχει η Ευρώπη να εντάσσεται στη μεταχείριση, σε αυτή τη μεταχείριση αυτών των ανθρώπων. Ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή μα είπε ότι υπάρχουν κάποιε οδηγίε σε ό,τι αφορά ε, τους δραστηριστέ ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά εκεί έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με προστασία, αλλά και με πρόληψη. Και γι' αυτό λοιπόν και έναντι των άλλων υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, δηλαδή να υπάρχουν κάποιε πρωτοβουλίε οι οποίε λαμβάνονται και από την πλευρά μα, να μεταβαίνουμε εκεί όταν υπάρχουν καταγγελίε και να τι ερευνούμε περαιτέρω. έχω να θέσω και ένα ερώτημα στον κύριο Κοβάλεφ Πώς αξιολογείτε εσείς ε, τη ρωσική δικαιοσύνη. Ε, προφανώς είναι δύσκολο να κινηθούν διαδικασίες κατά τέτοιων ομάδων ε, θανάτου, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, περιπτώσεις παραβάσεων. Τι θεωρείτε, είναι δυνατή μια μεταρρύθμιση αυτού του δικαστικού συστήματος ή όχι. Ε, και ένα ακόμα ζήτημα θα ήθελα να θέσω. Ε, σε σχέση και με τη διαδικασία διαβούλευση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία για την κοινωνία των πολιτών. Πώ αξιολογείται αυτό το νόμο ο οποίο υιοθετήθηκε πριν από μερικά χρόνια, ο οποίο προβλέπει ουσιαστικά περιορισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά τι ενέργειέ του. Ο πρώην πρόεδρο ε, Πούτιν είχε πει πώ ε, ο νόμο αυτό θα μεταρρυθμιστεί. Έγινε κάτι τέτοιο αποτελεί τελικά κάτι τέτοιο ένα εμπόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Εγώ έχω ε, να αναφερθώ σε κάτι ε, παλιό αν θέλετε που είναι οι διαβουλεύσεις, διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία. Ευρώπη δηλαδή και η Ρωσία σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων ως δύο διαφορετικοί πολιτισμοί. Για να τουλάχιστον εξετάσουμε το, ε, αυτή τη συζήτηση επίσημα επίπεδα. Συνεχίζονται λοιπόν διαβουλεύσεις, διμερείς διαβουλεύσεις, χωρίς αποτέλεσμα. Χαιρόμαστε που συνεχίζονται αυτές οι διαβουλεύσεις και θα συνεχίσουν στο διηνεκέ. Και εμεί βέβαια θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση. Επίσης αιώνιος. Ε, πολλές φορές αναφέρεται ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν ε, ανούσες συζητήσεις ε, σε σύγκριση με το να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε εδώ. Ε, δηλαδή, ε, ουσιαστικά ε, με τον τρόπο που κινούμαστε δεν ανταποκρινόμαστε τελικά στις δικές μας αρχές και ίσως αυτό να είναι τελικά ε, και ο στόχος ε, της Ρωσίας, δηλαδή να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ κοφών, αν θέλετε, δηλαδή από τις δύο πλευρές. Είμαστε ευχαριστημένοι με κάτι τέτοιο. Αυτό το ερώτημα το θέτω σε όλους μας. Όχι μόνο στους Ρώσους συναδέλφους μας. Γιατί εκείνοι δεν μπορούν να αποφασίσουν. Ακόμα κάτι μπορούμε να αποφασίσουμε και μέσα από την πλευρά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαντσμπέργκης. Ο κύριο Σούλτς. Ε, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τον ε, βαθύ σεβασμό μου απέναντι στους ε, υπέρμαχους εδώ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Εγώ ο ίδιος ήμουν δραστήριο στην αντιπολίτευση της λαϊκής δημοκρατίας της Γερμανίας και μπορώ να φανταστώ λίγο ε, πόσο πολιτικό, αν θέλετε, κουράγιο και θάρρος ε, πρέπει εσείς να έχετε ε, για να Κάντε αυτό που κάνετε σήμερα στη Ρωσία. Εμεί είχαμε, απειλούμασταν ε, με φυλάκιση από το καθεστώς τη τάση, δηλαδή τη πρώην ανατολική ε, Γερμανίας, αλλά εσά ε, εσείς απειλείστε με θάνατο, οπότε μπορώ να αντιληφθώ την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Όμω θα ήθελα να ακούσω λίγα από εσά σε ό,τι αφορά το ρόλο τη Ορθόδοξη Εκκλησία στη Ρωσία. Γιατί εμεί, για παράδειγμα, στην Πολωνία, στην Ανατολική Γερμανία, βλέπαμε να, την ε, βοήθεια της Ευαγγελικής Εκκλησίας ε, στην Ανατολική Γερμανία, της Καθολικής στην ε, Πολωνία. Ε, όμως διαπιστώνουμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Ρωσία ε, δεν παρέχει αυτή τη βοήθεια, δηλαδή συνεργάζεται με τον κρατικό μηχανισμό, παρότι θα ήταν ο, ο μοναδικός θεσμός ο οποίος θα μπορούσε να δράσει ε, κατά κάποιο τρόπο προ όφελο ε, των ε, διοκόμενων. Υπάρχει κάποιος ε, τρόπος για να αναλάβει αυτό το ρόλο η Εκκλησία. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους Ρώσους ευρωστεκλημένους μας. Ποιο θα ήθελε να παίρνει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εστιάσω στο ζήτημα της ε, ατομικής ευθύνης και της κρατικής ευθύνης. Κάτι τη διεξαγωγή της έρευνάς μας εστιάσαμε σε εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα αυτά και μιλάμε για ανθρώπους ε, με πολύ υψηλά αξιώματα μέσα στις ε, ρωσικές αρχές. Κανένας που ε, δεν θα πρέπει να παραμείνει ατιμόρυτος, αλλά υπάρχουν και πρόσωπα μέσα στις δομές εξουσίας, τα οποία δεν έχουν ε, διαπράξει τέτοια κλίματα με τα ίδια τους τα χέρια, αλλά και των οποίων η ευθύνη για αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν Κατά τη δική μας έρευνα, ε, εστιάσαμε σε ένα δίκλο ανθρώπων που θεωρούνται υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα. Ε, εάν λοιπόν ρίξετε μια ματιά στο κατάλογο αυτών των ονομάτων που περιλαμβάνεται στο δεύτερο τμήμα της μελέτης μας, θα δείτε πως ε, πολλοί από αυτούς είναι οι ομόλογοι σας στα διάφορα διεθνή φόρα. Εμείς λοιπόν διαθέσαμε ένα προκατακτικό κατάλογο αυτών των ονομάτων, αλλά η επιστολή μας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πως ε, εμείς ε, έχουμε πλέον διασφαλίσει πως ε, πράγματι βαρύνει ενοχή αυτά τα άτομα και ούτε και τα συγκεκριμένα εγκλήματα, λέγοντας πως θεωρούνται πως ε, θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνα, σημαίνει ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία εμείς ε, μπορέσαμε να συλλέξουμε και, τα, και στα οποία βασίσαμε την έρευνά μας, ε, μας οδήγησαν στο να, να έχουμε λόγους να πιστεύουμε πως τα εν λόγω άτομα είχαν εμπλακεί στην, στο να δοθεί η εντολή ή δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να αποτραπεί η διάπραξη του εν λόγω ερχόμενη σε αντίθεση με την δική την δημοσιασία. Και θεωρούμε ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν προσαχθεί ενώπιον της ποινική δικαιοσύνης. Ε, καθώς δεν έγιναν έρευνες, δεν ολοκληρώθηκαν έρευνες ή δεν έγιναν με αμερόληπτο τρόπο ή έγιναν με τρόπο ο οποίος ουσιαστικά να προστατεύει τους κατηγορούμενους από ποινική ευθύνη. Η αναφορά λοιπόν σε αυτή την υποτιθέμενη ενοχή αυτών των ατόμων δεν λέμε πως αυτά τα άτομα συμμετείχαν σε όλη την ουσιαστική δηλαδή διάπραξη του εγκλήματος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή η αυτουργία, η ευθύνη σχετίζεται με όλα, με όλους τους τρόπους όπω όπως αυτή καλύπτονται από το Διεθνέ ε, δίκαιο, ε, δηλαδή ο σχεδιασμός, η συμβολή στο σχεδιασμό ε, της διάπραξης ενό εγκλήματο, ατομικά ή από κοινού με άλλα πρόσωπα, με κοινό στόχο, και με κοινό σχέδιο, αλλά και η ευθύνη όπως αυτή βαρύνει του ανωτέρου. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην μελέτη μας στα, στις πηγές των στοιχείων που εμεί συλλέξαμε των αποδεικτικών στοιχείων και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρει και να δώσω έμφαση σε ένα τέταρτο. Καταρχήν στοιχεία από μη κυβερνητικέ οργανώσει, τα οποία σα έχουμε βέβαια διαβιβάσει και σε μεγάλε ποσότητε. Ε, δεύτερο, είναι αποφάσει ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι αποφάσεις αυτές πέρα από στοιχεία περιλαμβάνουν και παραπομπές σε πολύ σημαντικά έγγραφα τα οποία είχαν συνταχθεί σε εθνικό επίπεδο κατά την, ε, τις προκαταρτικές έρευνες και είχαν ε, ε, υποβληθεί από τις ρωσικές αρχές στην, στο δικαστήριο προς εξέταση και ένα τρίτο, μια τρίτη ομάδα στοιχείων τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά για να οδηγηθούμε στα συμπεράσματα της μελέτης μας. Έχουμε α, λοιπόν στη διάθεσή μας κάποιες, κάποια διατάγματα και κάποιες εντολές από πλευρά του Προέδρου Μεντεβέντεφ, ε, εγχειρίδια, ε, υπομνήματα, ε, φυλάδια και ό,τι καθεξής που αναφέρονται, αναφέρουν στοιχεία σε ό,τι αφορά τις ενόπλες δυνάμεις όπου αυτές έχουν ε, όπως ανα, κάνουν λόγο για την εμπειρία τους όπως και αναφέρουν και συγκεκριμένα ε, αξιώματα όπως αυτά κατέχονταν από, ε, από συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία σας τα υποβάλλουμε προς δική σας ε, για προκειμένου να τα εξετάσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Η κυρία Βιντάλ έχει το λόγο. Είναι η πρόσωπό μας από τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Γαλλικά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να αρχίσω θυμίζοντας ότι 22 δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στην άσκηση του έργου τους από το Μάρτιο του 2000 στη Ρωσία. Μία μόνο υπόθεση έχει διαλευκανθεί. Στις 7 Οκτωβρίου, συλλογισμένα στην τρίτη επέτειο της δολοφονίας της Πολιτόφσκα Γιάννα Πολιτόφσκα στη Μόσχα, κανένας ακόμα δεν έχει βρεθεί είτε εκτελεστής είτε ηθικός αυτούργος στη Ρωσία. Στην πρώτη δίκη ήταν κοινός ανάγκαμα έγινε σχετικά με τους υπεύθυνους και τους συνενόχους για την δολοφονία αυτής της δημοσιογράφου, η οποία δούλευε ειδικά για τον Κάφκασο. Μιλάμε λοιπόν για ατιμορρησία και η πλήρης είναι η ατιμορρησία όσον αφορά την πολιτική βία και αυτή η βία ασκείται σε βάρος όλων αυτών που επιχειρούν να διαδώσουν να μεταδώσουν πληροφορίες που δεν συμφωνούν με την, μια φυσιολογική, μια ψευδέστηση φυσιολογικής κατάστασης που προσπαθούν να παρουσιάσουν οι αρχές. Στον Κάφκας όμως, τι μας λένε, α, όλα επανήλθαν στο φυσιολογικό, δεν υπάρχει πια πόλεμος, φυσικά δεν υπάρχει ένοπλο κίνημα, αλλά έχουμε ένοπλο, συγγνώμη, εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος σοβεί και συνεχίζεται σιωπηλά. Πρόσφατα, στην Τσεσενία, στην στο Ντάγκεστάν πήγαμε να δούμε επί τόπου πώς δουλεύουν οι δημοσιογράφοι. Ε, λοιπόν, δεν υπάρχει ελεύθερο τύπο ούτε στη Τσετσενία ούτε στην Ιγκουσιτέα. Λίγο στην Τακιστάν. Δεν υπάρχει ελεύθερο τύπο. Υπάρχουν όμω προσπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσπαθούν να βοηθήσουν του δημοσιογράφου. Αντι, μάλλον αντικαθιστούν κατά κάποιο του δημοσιογράφου οι οποίοι είτε έφυγαν είτε δολοφονήθηκαν. Υπάρχει και ένα, στο Γκρόσνη ένα άγαλμα ε, για τους ε, δημοσιογράφους που πέθουν. Αυτό είναι όμως μια γούστου ηρωνία. Μερικούς που συναντήσαμε ξαφνικά άρχισαν να εξαφανίζονται. Η Εστεμίροβα, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ να κάνουμε αυτή την αποστολή και τις συνεντεύξεις, είναι νεκρή στην Τσετσενία. Άλλοι συνεχίζουν να πεθαίνουν. Και εμείς εδώ συζητάμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Σας ζητάω Σα ρωτάω συγκεκριμένα, είστε διευθυμένοι να πάτε στην Τσετσενία, στην Κουσεδία, στο Ταγκεστάν, να δώσετε βίζα σε αυτού που απειλούνται και που είναι εύκολο να ξέρετε ποιοι είναι. Είστε διευθυμένοι να, ε, να πληρώσετε για τη μετάφραση των μέσων ενημέρωση στι περιοχέ αυτέ, ώστε να μην έχουμε μια βιτρίνα του καθεστώτο. Αν είστε διευθυμένοι να το κάνετε αυτό, τότε είστε διευθυμένοι να του βοηθήσετε. Και αν θέλετε να του βοηθήσετε, τότε δεν είστε τελείω άχρηστοι. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Βιντάλ. Έχουμε ερωτήσει λοιπόν και προς την Κομισιόν και προς το Συμβούλιο. Θα ακούσουμε μετά. Συνεχίζουμε τον καταλογό μου. Έχω έναν συνάδελφο καταρχήν, τον κύριο Ντόνσκης. Θα του δώσω το λόγο και μετά Αντρέινε Κρασόφ. ο κύριος Κοβαλιόφ που έθεσε ερωτήματα και αυτός με στόχο να ακούσουμε τον κύριο Δημητριεύσκη αν εξακολουθούμε να έχουμε καλή επαφή και μετά η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Συνάδελφοι ευρωβουλευτές, αν θέλετε ζητήστε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση. Θυμάμαι παλιότερα οι διαφωνούντε και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους τρομοκρατούσαν, του ασκούσαν τρομερή πίεση, του στερούσαν πολλά, αλλά στη δεκαετία του 70 υπήρχε η δυνατότητα να κάποιο να απελαθεί από τη Σοβιετική Ένωση ή όπως ο Βλαμί Μπουκόφσκι να ανταλλαχτεί με τον Λουίς Κορβαλάν Φερρυπίν. Τώρα όμως στη Ρωσική Ομοσπονδία η κατάσταση έχει επιδεινωθεί αφόρητα αυτού του είδου οι δολοφονίες αντί για άλλε λύσει τις είχαμε ποτέ. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να μην ανεχτούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί αν ανεχτούμε ή τουλάχιστον σχετικοποιήσουμε πράγματα που έχουν σχέση με εγκληματική πολιτική και με απόλυτο κινησμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε μοιραζόμαστε την ευθύνη αυτή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το θάρρος των Ρώσων φίλων, αλλά πρέπει που πλέον να κάνουμε κάτι για να τους δοθεί η δυνατότητα να διαδώσουν τον καλό λόγο για το τι συμβαίνει στη Ρωσία και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατευτεί η ζωή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντόρσκι. Παρακαλώ τον κύριο Νεκράσοφ, ανεξάρτητο σκηνοθέτη, το οποίο το νέο φιλμ για τον πόλεμο Γεωργίας Ρωσίας στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ενίοτε είναι χρήσιμο να χρησιμοποιεί κανείς απλή γλώσσα. Θα έρθω σε αυτό που ανάφερε ο κύριος Λαντσμπέργης. Λόγια και κούφια λόγια. Νομίζω υπάρχει μια βασική αντίφαση. Σε αυτό που εγώ θα το πω διασυνοριακή δικαιοδοσία Αυτό που θεωρεί η Ένωση και οι διεθνείς οργανισμοί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν διασυνοριακά. Κάποιος παραβιάζει τα δικαιώματα με πολιτικές δολοφονίες κλπ. Σοβαρές δηλαδή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ακούσαμε. Δεν πρέπει να θεωρηθούν μόνο της δικαιοδοσίας μόνο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ωστόσο όλοι ξέρουμε την καταστολή την δίωξη μη κυβερνητικών οργανώσεων με, στη Ρωσία με στόχο να στερηθούν τα υλικά μέσα, λεφτά με άλλα λόγια, προκειμένου να λειτουργούν. Το λέμε αυτό κινησμό εκ μέρους της ρωσικής κυβέρνησης. Πέστε το όπως θέλετε, αλλά είναι κάτι πολύ πολύ πρακτικό. Δεν μετράει η ιδεολογία σήμερα δεν μιλάνε τα ωραία λόγια. Είναι κάτι που κάνει ζημιά. Δράση και λεφτά. Αυτό κάνει ζημιά. Συμφωνώ με τον προλαγίσαντα Αναφερθήκατε στον κύριο Μουράτοφ. Ίσως ο κύριος Μουράτοφ να μην χρειάζεται λεφτά γιατί η εφημερίδα του λειτουργεί εμπορικά. Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ξοδεύουν την τελευταία τους δεκάρα και μερικές φορές δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους προκειμένου να δημοσιεύσουν μία σελίδα μια εφημερίδα μια σελίδα που την κάνουν μόνοι τους στις επαρχίες και στο Σεν Πέτερσπουργκ από το οποίο προέρχομαι χρειάζονται λεφτά και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε να φοιτητές λοιπά να έρθουν εδώ. Πολύ σημαντικό αυτό, εξελικτικά θα βοηθήσει, αλλά υπάρχουν πολύ πιο επίγοντα ερωτήματα και προβλήματα. Τι μπορεί να γίνει σήμερα ή χθε θα έλεγα, πριν είναι πολύ αργά. Ελπίζω αυτή η αντίφαση ανάμεσα στην ε, θεωρητική διασυνορική ισχύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την βούληση όλων να βοηθήσουν μπορεί να επιληθεί με έναν πρακτικό τρόπο. Μεταξύ άλλων, η ρεαλιστική πρόθεση στην πληθώρα αυτών των νόμων που βγάζει η Ρωσική Ομοσπονδία προκειμένου να κόψει τη ροή μέσων για βοήθεια των στελεχών που δουλεύουν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ακτιβιστών. Εγώ προέρχομαι από τον κύκλο των δημοσιογράφων και των σκηνοθετών και επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι η ελευθερία πληροφόρησης, η ελευθερία λόγου είναι ένα από τα θεμελιώδη δεδομένα προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση στη Ρωσία. Όχι μόνο η ελίτ που έχει τη δυνατότητα να βγάλει ένα διαβατήριο και να έρθει εδώ οι φοιτητέ, αλλά ο μέσο Ρώσο είναι πολύ ευαίσθητο Πολλοί άνθρωποι είναι ευγενείς άνθρωποι που στερούνται της πληροφορίας και υφίστανται πλήση εγκεφάλου. Περάστε αυτή την πληροφορία, σπάστε αυτό το σιδηρού παραπέτασμα που υπάρχει. Πολλοί δημοσιογράφοι εδώ, με οργανώσεις και πολιτικοί, μπορείτε να συνεργαστείτε και με αυτούς. Σπάστε αυτό το σιδηρού παραπέτασμα που εμποδίζει την κίνηση της πληροφορίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, αυτό ακριβώς καταλαβαίνουμε που λέτε ότι υπάρχει ένα σιδερούν ε, παραπέτασμα που πρέπει να σπάσουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Να συνεχίσω μετά από τον κύριο Λάνκες για το θέμα των διαβουλεύσεων, του διαλόγου που συνεχίζεται η ΣΑΗ. Συναντήσεις σαν και αυτήν που είχαμε σήμερα είναι συναντήσεις σημαντικές για μας. Μας δίνουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ακούσουμε αυθεντική ενημέρωση από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μια σκληρή πραγματικότητα στη Ρωσία, αλλά και σε άλλα σημεία του κόσμου. Πάντως, πρέπει να πω ότι είμαι κάπως απεσιόδοξος. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά σαν ρουτίνα. Δηλαδή, μετά τη σημερινή συζήτηση θα πούμε στους αυτούς μας ωραία, είχαμε ανοιχτό διάλογο με τους φίλους μας από τη Ρωσία. Και αυτό ήτανε. Όχι, κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν αλλάζει η ζωή μας από τη μια στιγμή στην άλλη. Μερικές φορές χρειάζεται πίεση για πολύ χρόνο και μόνο τότε φαίνεται κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε εμείς, η Κομισιόν, το Συμβούλιο, η Σουδική Προεδρία δεν πρέπει να νιώθουμε ευχαριστημένοι επειδή ναι, έχουμε αυτές τις διαβουλεύσεις με τη Ρωσία. Μπορεί κανείς να είναι θετικός για αυτές, αλλά δεν πρέπει αυτό να φτάνει. Γι' αυτό λοιπόν και χαίρομαι που άκουσα κάποιον να λέει ότι στην νικουσία θα πάει πήγε μάλλον μια αποστολή, πήγανε, ήπιανε τζάι με τον πρόεδρο και γύρισαν και είπαν τι ωραία που συζητήσαμε. Μα ακριβώ αυτό είναι που πρέπει εμείς να αποφύγουμε, να μην γίνεται αυτό και εδώ, να μην μας ικανοποιεί αυτό. Εγώ δεν έχω ειδική πρόταση εδώ για να σας πω πώς θα μπορούσαμε να πιέσουμε την κατάσταση ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Μπορώ όμως να σας πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε τι είναι αυτό το κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε εκτός από αυτές τις ε, συναντήσεις. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους Ρώσους προσκεκλημένους μας. Ακούγοντας τον ε, Σιγκεργέη Κοβαλιεφ πριν από λίγο καιρό, μου φάνηκε ότι υπήρχε μια αλήθεια σε αυτά που είπατε τότε, ότι κάτι θα άλλαζε, σε βάθος θα άλλαζε ήταν ακριβώς η στιγμή που είχαμε την πρώτη σύραξη στην Τσετσενία. Τότε δηλαδή που αναρωτηθήκαμε μήπως η Ρωσία ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έπρεπε να σταματήσει να είναι μέλος. Και τότε μας είχατε πει ότι μα πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία γιατί αν δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος σε διεθνές επίπεδα τότε θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ότι θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε έναν τρόπο να προκαλούμε τις αλλαγές. Σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα, πρέπει να σας πω ότι τα λόγια σας, κυρίες και κύριοι, μας εντυπωσίασαν πάρα πολύ. Καθημερινά ενημερωνόμαστε από διάφορες πλευρές για τα πράγματα που συμβαίνουν, είτε με τους δημοσιογράφους, είτε με αγωνιστές, είτε με μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλους που θέλουν να υπογραμμίσουν τη σημασία που έχουν τα έθνη, όπως την Τσετσένια. Όλα αυτά είναι εντυπωσιακά, αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνουμε πλήρως τι σημαίνει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει ένα σωρό προβλήματα τα οποία μας υπεβεβαιώσατε και σήμερα με τις παρεμβάσεις σας και την παρουσία σας εδώ. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως την αποφασιστικότητά σας. Έχει να κάνει με το ότι θα θέλατε να ευαισθητοποιήσετε το σώμα. Να μην είναι μόνο ένα κοινοβούλιο ανθρώπων ε, που συνεδριάζουν σε επιτροπές, εξάλλου υπάρχουν και άλλα όργανα πιο σημαντικά από το Κοινοβούλιο, αλλά εσείς αυτό που θέλετε είναι όλοι εμείς να μην ξεχάσουμε. Επειδή υπάρχει κρίση, προβλήματα με την ασφάλεια, ενέργεια κτλ. Να μην ξεχνάμε την ίδια την ουσία της λειτουργίας ενός κράτους. Η ουσία λειτουργίας ενός κράτους είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών ότι αυτό είναι το θεμελιώδες και ότι αυτό πρέπει να παραμείνει, να μην το ξεχνάμε και να φροντίσουμε σε αυτούς που είναι τέροι μας, γείτονές μας, να τους το δείξουμε, να φροντίσουμε να δεχτούν αυτές τις προδιαγραφές που είναι τόσο σημαντικές για μας και να φροντίσουν να τις σέβονται. Έχουμε εμπειρίε με διάφορους γείτονε για θέματα που έχουν να κάνουν εδώ και 70 χρόνια που δύσκολα μπορεί κανείς σήμερα να εξηγήσει. Εμείς που βρισκόμαστε και δίπλα φτιάξαμε μια επιτροπή Πολωνίας-Ρωσίας με εμπειρογνώμονες ώστε να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια προβλήματα. Και γι' αυτό ακριβώς καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να συζητήσει κανείς για επίκαιρα θέματα, για σύγχρονα όσοι συμμετείχαν στο παρελθόν σε όλες αυτές τις ιστορίες που σκότωσαν πολωνούς αξιωματούχου, για παράδειγμα δεν υπάρχουν πια στη ζωή αλλά όταν πρόκειται για σύγχρονα γεγονότα που οι υπεύθυνοι είναι μεταξύ μα, εκείνοι που έχουν δώσει την εντολή για τις δολοφονίες για παράδειγμα τότε είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Όμως παρόλα αυτά είναι χρέος μας να μην μείνουμε παρατηρητές να δράσουμε. Οι δραστηριότητές μας πρέπει να είναι τέτοιες που να υπενθυμίζουν συνεχώς τις αξίες που πρέπει να τηρούνται. Και υπάρχουν διαφορετικοί χώροι, διαφορετικά φόρα στα οποία πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζουμε αυτές τις αρχές. Να μην είναι αυτό ο στόχος, το τελευταίο, να είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο θα φτιάξουμε την κοινωνία και εκείνη της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, σεβόμενη την ιστορία, τόσο δύσκολη, περίπλοκη αυτής της χώρας. Ξέρουμε τι έγινε εκεί. Αλλά πρέπει να σεβόμαστε και τις αρχές που σέβονται τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι αρχές πρέπει να εφαρμόζονται η ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Λαντσμπέργης νομίζω ότι πολύ καλά το περιέγραψε. Έτσι πολύ συμπυκνωμένα, αλλά τόσο σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρίψη. Ο Αντιπρόεδρος Καζάκη, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Θέλω και εγώ να μεταφέρω την εντύπωση που μου έκαναν τα λόγια σας και οι παρεμβάσεις σας. Θυμήθηκα τα τελευταία γεγονότα στις χώρες μας, τέως ε, σοβιετικό μπλοκ η χώρα η οποία προκάλεσε ε, την καταστροφή του σιδηρού πετάσματος που έφερε τη δημοκρατία στις χώρες μας τέος Σοβιετικού μπλοκ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία κλπ. Ήταν ακριβώς η Ρωσία. Από την Ρωσία ξεκίνησε η Γκλάσνοστ, η διαφάνεια, η περεστρόικα. Και όλα αυτά οδήγησαν σε μια σε ένα πλήρη δημοκρατισμό και στο γεγονός ότι η Βουλγαρία και οι άλλες χώρες τέος στο Σοβιετικό μπλοκ εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδοξο είναι ότι η χώρα η οποία προκάλεσε όλες αυτές τις αλλαγές σήμερα διαπιστώνουμε ότι επιστρέφει στον ολοκληρωτισμό, στην έλλειψη ελευθερίας σκέψης και λόγου. Μια χώρα όπου οι άνθρωποι διώκονται εξαιτία των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια μεγάλη χώρα και μια μεγάλη δύναμη έχει σαν αποτέλεσμα όλες οι υπόλοιπες χώρες να είναι επιφυλακτικές απέναντί τους, επιφυλακτικές να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, να ενοχλήσουν περισσότερο αυτή τη χώρα. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, τον κύριο Τίμανς τόσα μας είπε και τελικά κατέληξε το συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να μπορεί να επιβάλλει τις διεκδικήσεις της στη Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εννοείται ότι τα οικονομικά συμφέροντα και άλλα, οι σχέσεις μας εμπορικές και οικονομικές με τη Ρωσία είναι πάρα πολύ σημαντικές για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ως υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν δράσουμε με... σε συνεργασία με άλλες με άλλους οργανισμούς όπου συμμετέχει και η Ρωσία, Συμβούλιο της Ευρώπης για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν και όλες οι δομές του ΟΗΕ, ο ΑΣΕ, όπου η Ρωσία συμμετέχει. Αν λοιπόν εμείς συνεργαστούμε πιο στενά με όλους αυτούς και θέτουμε συνεχώς το θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ίδια ένταση και στο ίδιο μήκο κύματο, τότε πιστεύω ότι θα μπορούμε να ασκήσουμε πίεση και επιρροή γιατί στο κάτω-κάτω η Ρωσία δεν μπορεί να απομονωθεί, δεν μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό και σας συγχαίρω για τις πρωτοβουλίες σας, ε, κυρία Πρόεδρε, για τη συνάντησή σας με τον αρμόδιο για ανθρώπινα δικαιώματα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι ο σωστός δρόμος για να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε Καζάκ. Φίξατε το ζήτημα των χωρών αυτών που γεννήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση πριν από 20 χρόνια και υπάρχουν και άλλες χώρες που παρέμειναν φυλακισμένες. Οι υπηρεσίες ασφάλειας, τους σκότους όμως δεν διαλύθηκαν, δεν είδαν το φως. Είναι ακριβώς το κίνημα, να, ο κύριος Σούλς μίλησε για την Τέσσερα Ανατολική Γερμανία, το κίνημα αυτό επιτάχυνε την κατάσταση. Αυτό ακριβώς είναι που έπρεπε να γίνει το 1991. Έγινε στο Βερολίνο, αλλού όμως ποτέ στη Ρωσία Σοβιετική Ένωση. Θα δώσω την ευκαιρία στους συναδέρφους να πάρουν το λόγο πάλι και θα ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Θέλω να σας πω ότι μεταξύ των συμμετοχόντων υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη Ρωσία. Ε, μέλη της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αν και εσείς θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Μπορείτε. Ο κύριος Τόκης τώρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν ιδιαίτερα τον κύριο Κοβάλεφ και τους υπόλοιπους Ρώσους προσκεκλισμένους μας και να τους ε, καλωσορίσω εδώ. Ε, Είστε πολύ ευπρόσδεκτοι και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε ότι θα πρέπει επιτέλους να δράσουμε, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να μιλάμε πλέον. Εγώ ταράχθηκα χθε όταν άκουσα στην ε, τηλεόραση ότι κατέστη πλέον σαφές ότι η Μαργαρέτη Σφέτσερ και άλλοι ε, και άλλες ηγετικές πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης ήταν κατά της ε, κατάρρευσης ε, του τείχους και οι πολιτικές αυτές προσωπικότητες έκαναν, προέβησαν σε διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά με αυτό το σκεπτικό. Και τα εν λόγω αρχεία ανοίχθηκαν πλέον και είναι πλέον διαθέσιμα τα λόγω έγγραφα και ήρθαν στο φως της ε, δημοσιότητας. Εγώ έρχομαι από τη Ρουμανία και ε, θυμήθηκα πολλά πράγματα Ε, το Υπουδαπέστη του 56, Ζολιντανός και της ε, Πολωνίας και ούτω καθεξής τέτοιες κινήσεις δηλαδή οι οποίες ε, χαιρετίστηκαν από την Ευρώπη, άνθρωποι όπως ο Ζαχάροφ έλαβαν εκτίμηση και κύρος για το θάρρος τους, αλλά ταυτόχρονα είχε ασκηθεί και μια πολιτική υπερδυνάμεων η οποία ουσιαστικά υποτιμούσε αυτές τις αρχές, δηλαδή τις αρχές της δημοκρατίας, ε, του κράτους δικαίου, γενικά δηλαδή τις βασικές ηθικές αξίες της δύση. Μερικές φορές λοιπόν δεν δίνονταν προτεραιότητα σε αυτές τις αρχές. Εγώ ε, κατά τις δεκαετίες του 70 και του 80 ήμουν ιερέας, μετά είναι και επίσκοπος και δεν θα ξεχάσω όσο πολύ έπρεπε να αγωνιστούμε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και στην παγκόσμια διάστηση της Λουθυρανικής Εκκλησίας κατά της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας καθώς ε, ε, πολλοί ιερείς ε, του μετακομμουνιστικού καθεστώτος σε αυτές τις οργανώσεις ε, συνεργάζονταν με τα κομμουνιστικά καθεστώτα, μερικέ φορέ μάλιστα και με τι υπηρεσίες ασφαλείας. Και μάλιστα ένα τέτοιο άτομο ήταν και επικεφαλής της ε, Παγκόσμιας ε, Ένωσης της Εκκλησίας των Μεταρρυθμιστών και προσπαθούσε βέβαια πάντα να καταπιέσει ανθρώπους όπως εμένα εμείς βέβαια προσπαθήσαμε πάντοτε να τον ε, πολεμήσουμε και είχαμε και το θάρρος να αντιταχθούμε ανοιχτά σε αυτόν και στα καθεστώτα αυτά. Και δυστυχώς ε, εξακολουθώ να διαστάνομαι αυτό το διπρόσωπο, αν θέλετε, χαρακτήρα Δηλαδή από τη μία πλευρά γνωρίζουμε τα όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωση, στις διάφορες διασκέψεις, στα διάφορα φόρα, όπου συγχαίρουμε αυτούς τους ανθρώπους για το θάρρος και το κουράγιο, και το κουράγιο τους, αλλά από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι οι δυτικές χώρες, οι βιομηχανικές χώρες, διστάζουν ε, πολύ να ε, λάβουν μέτρα Ε, αυτό νομίζω πως αποτελεί ένα κληροδότημα του παρελθόντος, αλλά θα πρέπει επιτέλους να το εγκαταλείψουμε. Ωραία είναι να λέμε εδώ τόσο μακριά από πράγματα για το Θιβέτ, ε, για τους ε, Ουιγούρους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε βέβαια και την ενεργειακή πολιτική με τη Ρωσία, που σημαίνουν δηλαδή ότι έχουμε και οικονομικά συμφέροντα. Αυτά θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Τέτοιου είδου συμφέροντα όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα δικαιώματα και με ελευθερία. Εγώ είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που μπορώ να είμαι μέλος αυτής της ε, Επιτροπής η οποία δηλαδή ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζω να καταστεί ε, δυνατόν κάποια στιγμή στο μέλλον να υπάρχει ένα αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενός δηλαδή επιτετραμένου, ο οποίος ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο οποίος θα μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται και εκτός Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τούκες για την παρέμβασή σας. Νομίζω πως ε, θα ήταν ε, τώρα σωστή χρονική στιγμή αν θα ήθελε να συμμετάσχει στη συζήτησή μας στο Στάνισλαβ Δημητριεύστη έχουμε ακόμα αυτή τη σύνδεση. Υπάρχει. Ίσως πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ίσως θα μπορούσε να πάρει κανείς το λόγο και μετά. Α, να του δώσουμε το λόγο. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους προσκεκριμένους μας για τις μαρτυρίες τους, όσα μας είπαν. Επίσης, θέλω να εκφράσω και το θαυμασμό μου για το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους. Αμέσως θέλω να πω για την πρόσκληση που μας έκανε εκπρόσωπος των Reporters χωρίς ε, σύνορα, το δημοσιογράφο χωρίς σύνορα. Μας πρόσφερε διάφορες προσκλήσεις, έκανε διάφορες προτάσεις. Η απάντησή μου είναι ναι σε όλες. Και θα επιμείνω στην αναγκαιότητα όλοι αυτοί που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, θα πρέπει να προστατεύονται ή τέλο πάντων να μπορούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να μπορούν να χαίρουν θεωρήσεων από τις χώρες μας, ώστε να έχουν την δυνατότητα να μπορούν αν μη τι άλλο, να έχουν άμεση προστασία εφόσον αυτή χρειάζεται. Σήμερα με τις πληροφορίες, με τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτουμε, οι πρεσβείες μας μπορούν πολύ γρήγορα να ενημερωθούν για τους κινδύνους που υπάρχουν και έτσι να μπορούμε πολύ συγκεκριμένα να προσφέρουμε αυτή την προστασία. Θέλω να πω και δύο λόγια τώρα για το σκεπτικισμό που επικρατεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος εχθρός πιο επικίνδυνος για αυτούς που αγωνίζονται επί τόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το σκεπτικισμό. Έχω τον κύριο Τόκης εδώ, ο οποίος ε, μίλησε πριν από μένα και θυμάμαι τότε που ήταν στην ε, αντιπολίτευση στη χώρα μου στη Ρουμανία μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ εμείς που δεν είχαμε το θάρρος να κάνουμε ό,τι έκανε εκείνος, αυτός αποτέλεσε το παράδειγμα για μας. Καταλάβαμε ότι υπήρχαν ε, εκτός Ρουμανίας άνθρωποι οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να δώσουν αυτό τον αγώνα. Και έτσι μόνο με μια αισιοδοξία μπορούμε να κερδίσουμε. Ο σκεπτικισμός λοιπόν σίγουρα δεν είναι καλός σύμβουλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρέντα, λοιπόν βλέπω ότι έχουμε την σύνδεση Skype με τον Στάνισλαβ Δημητρίευσκη. Λοιπόν, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την σημερινή συζήτηση εδώ. Έχετε σχόλια, θέλετε ίσως να κάνετε διευκρινήσεις, να μας πείτε τι μέτρα θα επιθυμούσατε να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακολούθησα πάρα πολύ καλά όλες τις παρεμβάσεις σας και ευχαριστώ και αυτούς φρόντισαν για τη σύνδεση Skype. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο απαιτητικοί και πιο επικριτικοί απέναντι στη Ρωσία. Μιλάτε για διαπραγματεύσεις με τη, Ρουσία, με τη Ρωσία, ναι. Σήμερα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κοινοτικά όργανα ζήτησαν από τις ρωσικές αρχές να ερευνήσουν τις δολοφονίες στην Τσενία, τις δολοφονίες αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ομοσπονδία ανταποκρίνεται σε τέτοιες, ε, τέτοια τίματα Λένε ναι, ναι, βεβαίως θα ερευνήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό λέει η Ρωσική Ομοσπονδία. Όμως ψεύδονται οι Ρώσοι αρμόδιοι ψεύδονται. Οι εκπρόσωποι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα γίνει ποτέ καμία έρευνα. Εδώ και χρόνια δεν έχει γίνει, ούτε θα γίνει ποτέ. Η Ρωσική Ομοσπονδία καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι οι εταίροι της γνωρίζουν επίσης πάρα πολύ καλά ότι ποτέ δεν θα γίνει τίποτα. Όλοι λοιπόν παριστάνουν, υποκρίνονται ότι καταλαβαίνουν κάτι άλλο και αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Εκερός είναι να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Σε λίγες εβδομάδες θα μιλήσω με αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τον κύριο Μεμπέργκ που είναι ο αρμόδιος ε, επιτεταμένος για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ζητήσαμε, του ζητήσαμε όταν πάει στη Τσετσενία να μην συναντήσει θύματα ε, στην επικράτεια του Κάντερεφ. Ότι έτσι καλλιώς δεν θα του πούνε την αλήθεια, ότι οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται και δεν θα μιλήσουν. Νομίζω ότι το κατάλαβε Πήγε όμως, αυτό έγινε νωρίτερα, πήγε λοιπόν και τα αποτελέσματα ήταν γνωστά. Οι συνάδελφοι μου είπαν ότι ο κύριος Μεβέρκ προσκλήθηκε από τον κύριο κατερόφ να πάει και δέχτηκε την πρόσκληση. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν ότι τέτοιες συναντήσεις με επίσημο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να προσκαλείς κάποιο σε δείπνο στον Κάφκασο. Αυτό είναι μια χειρονομία πολύ ιδιαίτερη. Αφήνεις δηλαδή κάποιον να μπει στο προσωπικό σου χώρο. Για μένα αυτή η χειρονομία είναι απαράδεκτη. Ο κύριος Καντερόφ προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να φτιάξει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς στην ε, Τσετσενία. Η Ρωσία στρέφεται, είπατε, προς την, ε, στον ολοκληρωτισμό. Ε, λοιπόν, η Τσιζενία είναι ε, ένα, ένας δακτύλιος μέσα σε αυτό όλο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ο εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν τον έχει συλλάβει, ενώ έχει ένα ορολόγος να το συλλάβει και να το καταδικάσει. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά καθίστε και σκεφτείτε το θέμα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί μια λύση. Όμως πρέπει να βρεθούν άλλα μέσα για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση που χειροτερεύει ολοταχώς. Για άλλη μια φορά ζητάω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτεί τη δημιουργία μιας ερευνητικής επιτροπής για τα διεθνή εγκλήματα που έλαβαν χώρα στον Βόρειο Κάφκασο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ Στάνισλαβ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Νομίζω ο κύριος Πρέντα και άλλοι θα να πάνε στην Γκουσέτια και στις άλλες περιοχές του Βόρειου Καυκάσου θα μπορούσαν και άλλοι να πάρουν μέρο σε αυτή την αποστολή και φυσικά να συνεργαστούμε με μη κυβερνητικέ οργανώσει και να συζητήσουμε και του εκπροσώπου τη Ρωσία. Αυτό που ήθελα να πω αυτή τη στιγμή είναι ο διπλωματικός εκπρόσωπο τη Ρωσία. παραπονέθηκε γιατί δεν τον προσκαλέσαμε. Προσκαλέσαμε όμως ένα εκπρόσωπο της Ρωσίας στη σημερινή μας συνεδρίαση. Με επέκρινε δρυμαίως. Είπε ότι ε, μεροληπτούμε έναντι της Ρωσίας και ενώ δεν μιλάμε για την Κίνα ή για άλλες χώρες πολλοί πρεσβευτές παραπονιόνται και λένε ότι ασχολείστε υπερβολικά με μας και ο πρεσβευτής ο ίδιος της Κίνας απάντησε σε μια πρόσκληση που του έστειλα στο παρελθόν ήρθε η στιγμή να ξαναδώσει το λόγο στον κύριο Κοβαλιόφ για να απαντήσει στα ερωτήματα που ετέθησαν παραδείγματος για το πρόγραμμα ανταλλαγών και πολλά άλλα ερωτήματα. Κύριε Κοβαλιόφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Κάρτερ, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, είπε κάτι εξαιρετικό. Είπε «Δεν μπορώ να στείλω τους πεζοναύτες για να απελευθερώσουν τους αντιρρησίες συνείδησης της Ρωσίας που είναι κρατούμενοι. Όλα τα άλλα μπορώ να τα κάνω». Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα περί του πρακτέου. Ένας άλλος σπουδαίος άνθρωπος, ο Ανδρέης Ζαχάροφ, τον Ιανουάριο του 88 είπε «Η χώρα μου χρειάζεται υποστήριξη αλλά και πίεση». Πιστεύω ότι πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο αυτή τη φράση σήμερα. Πρέπει να πούμε όχι μόνο η χώρα μου χρειάζεται υποστήριξη και πίεση, αλλά όλος ο κόσμος πρέπει να ασκήσει πίεση στη Ρωσία. Το πιστεύω αυτό απόλυτα. Τώρα, τι είδους πίεση. Δηλαδή, πώς πρέπει να δράσει κανείς. Εσείς, πεπειραμένοι πολιτικοί, ξέρετε πολύ καλύτερα ποια είναι η πιο κατάλληλη μορφή Άσκηση πολιτικής πίεσης. Αν μου ζητήσετε όμω τη συμβουλή μου, θα σα έλεγα ότι πρόσφατα το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε ένα ψήφισμα. Αναφέρθηκα σε αυτό πριν. Σύσταση στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να απευθυνθούν, να προσφύγουν μάλλον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ρωσίας. Κατά της Ρωσίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη υπέστη μια τέτοια προσφυγή και αποδέχτηκε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμορφώθηκε με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι, όλες οι χώρες αυτές εκπροσωπούνται από ευρωβουλευτές. Γιατί δεν μπορείτε να ζητήσετε από τις χώρες σας να εφαρμόσουν αυτό το ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι χώρες σας είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και κάτι άλλο. Εδώ μας δίνεται χρόνο μιλίας 6 με 10 λεπτά και αρχίζουμε να μιλάμε πολύ συγκίνηση. Εσείς που είστε εμπειρογνώμονες στην Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εσείς θα έπρεπε να γνωρίζετε σε βάθος το θέμα προκειμένου να κρίνετε ως εμπειρογνώμονες και να έχετε απόδειξη των κατηγοριών που εμείς σας παρουσιάζουμε. Γιατί δεν οργανώνετε ένα σεμινάριο για τους ευρωβουλευτές. Εγώ είμαι διατεθειμένος να μιλήσω και μία και δύο ώρες όπου θα είχα την ευκαιρία να πάω σε βάθος. Σε δέκα λεπτά δεν έχει νόημα. Άλλο. Αναφέρθηκα στο ερώτημα τι να κάνουμε και επίσης το ερώτημα εξίσου σημαντικό τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ε, λοιπόν, δεν πρέπει να πιστεύουμε αυτά που λένε οι επίσημοι εκπρόσωποι. Όλοι λένε ψέματα. Και είναι εύκολο αυτό να αποδειχθεί. Κυρίως δεν πρέπει να υποτασσόμαστε στη βλακώδη αρχή του πολιτικά ορθού. Το πολιτικά ορθόν θα είναι αυτό που αποκαλούμε επικυρίαρχη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι δημοκρατία, τελειώνει και παύλα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κυριαρχούσα δημοκρατία ή επικυρίαρχη δημοκρατία. Τι δεν πρέπει να κάνουμε, τι άλλο δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να λέμε συγχαρητήρια για υποτίθεται δημοκρατικές εκλογές. Και όλοι το κάνατε αυτό είναι του κυρίου Μεντβέντεφ. Τι είδους ελεκτές κέρδισαν αυτοί οι δύο. Εγώ, αν ήμουν επίσημος εκπρόσωπος μιας δυτικής χώρας, θα έλεγα το εξή στον κύριο Μετβέντεφ. Αγαπητέ μου κύριε Μεντβέντεφ, φυσικά δεν πρόκειται να κόψουμε τις σχέσεις με σας, την οικονομική μας συνεργασία κτλ. Αλλά εγώ ξέρω και εσείς το ξέρετε και οι δυο μας το ξέρουμε καλά ότι δεν είστε νόμιμος εκπρόσωπος, κάθε άλλο. Δεν είστε νόμιμος ηγέτης της χώρας σας. Γιατί σε μια δημοκρατική χώρα μόνο οι πολιτικοί ηγέτες που εκλέγονται άμεσα και δημοκρατικά θεωρούνται νόμιμοι εκπρόσωποι που να έχουν εκλεγεί από την ελεύθερη βούληση των εκλογέων. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με εσάς. Δεν σε συγχαίρω λοιπόν. Για το ότι υποτίθεται κερδίσετε αυτές τις εκλογές. Ας προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τις σχέσεις μας στην αλήθεια, στο αληθές. Αν ένας δυτικός ηγέτης έκανε κάτι τέτοιο, θα πετύχαινε προς έκπληξή του αποτελέσματα. Φυσικά και κατηγορίες και ε, κριτική, ε, ασκώντας κριτική κατά της ρωσικής ηγεσίας. Έπειτα μιλάμε για κρίση, ενεργειακή κρίση κλπ. Σα θυμίζω λοιπόν ότι αυτή η κρίση δεν είναι καινούριο φρούτο. Η πετρελαϊκή κρίση, πολλές τέτοιες κρίσεις έχει γνωρίσει ο κόσμος ως τώρα. Όταν η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να πάρει θέση στη Μέση Ανατολή, τότε η Δύση γνώρισε δύσκολες στιγμές Έκανε εξωπρεπείς προσπάθειες βέβαια η Δύση ξέρετε ένα εμπόρευμα έχει αξία μόνο αν μπορεί κανείς να το αγοράσει. Το πετρέλαιο δεν μπορεί κανείς ούτε να το πιει, μπορεί μόνο να το αγοράσει και να το πουλήσει και να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την πώλησή του για να αγοράσει τρόφιμα πούμε, να φάει. λέμε ότι πάει ο ψυχρός πόλεμος. Ξεχνάμε όμως ότι ο ψυχρός πόλεμος μερικοί τον έχασαν τον πόλεμο αυτό. Το ξεχνάμε. Ξαναγυρίζω στις δύο ερωτήσει μου. Τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Υπήρξε μια ερώτηση για την Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας συμμετέχει στη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς συμμετέχει. Ως εκκλησία. που είχε σχέσεις με τον κύριο Στάλιν και θυμάμαι πολύ παλιότερα Κάποιο μου έφερε ένα έγγραφο που είχε βρει σε μια εκκλησία, ένα, ένα χαρτί ήταν, που έλεγε, που ήταν γραμμένο στο χαρτί αυτό, ότι ζητούσαν αυτοί που έχουν αντικαθεστατικά έγραφα και κείμενα να δοθούν στους επικεφαλείς της Εκκλησίας. Αυτά έγραφε αυτό το χαρτί. Αυτά για την περίφημη αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ξέρετε ότι ένας από τους Ρώσους Πατριάρχες ήταν κατάσκοπος, πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ με το ψευδόνιμο Drogdov Αυτό έχει αποδειχθεί και κανένας δεν το διέψευσε. Συνεπώς η Εκκλησία πάντα ανα, ανακατευόταν στην ε, πολιτική ζωή και οι χριστιανοί παρόντες δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Κοβαλιόφ. Ακούσαμε πολλά σοφά λόγια. Θα προτιμούσα να είχατε περισσότερο χρόνο να μας μιλάτε, αλλά Ήρθε η ώρα τώρα να περάσουμε στην Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ας αρχίσουμε τον προσδευτή Νορλάντερ για να κλείσουμε το θέμα αυτό πρώτης, ε, ευρωπαϊκής, ε, πρώτης διάσκεψης κορυφής. Θα είμαι σύντομη κυρία Πρόεδρε. Και επειδή πρέπει να προλάβω την πτήση μου. Α, θα είμαι εκτό άλλου σύντομο. Ε, μαζί λοιπόν με αυτές τις συζητήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να λάβουμε και παράλληλα μέτρα. Ε, Προφανώ και υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι μουσιογράφοι και ούτω καθεστώ χρήζουν πρακτική αρρωγή επί τόπου. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ασκηθούν και πολιτικέ ή διπλωματικέ πιέσει. Γιατί αν δεν ασκηθούν αυτέ οι πιέσει, δεν μπορούμε να μπούμε στη Ρωσία για να παράσχουμε αυτή την πρακτική βοήθεια. Ε, και έτσι υπέρμαχοι των πολιτικών ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα μπορούν να καταλήψουν τη χώρα γιατί δεν θα αναβάνουν θεωρήσει και ούτω καθεξή. Προφανώ και οι κυβερνήσει έχουν να παίξουν διαφορετικό ρόλο από, τις, ε, από την κοινωνία των πολιτών. Εάν οι κυβερνήσει ε, προβούν σε μποϊκοτάζ ενό καθεστώτο ή κάνουν κάτι παρόμοιο, δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να επηρεάζουν το λόγο καθεστώ. Εάν όμως μη κυβερνητικέ οργανώσει δεν προβούν σε μποϊκοτάζ, τότε βέβαια δεν έχουν ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή του για να επιτύχουν του στόχου του. Επίση, να πω πω ε, ε, εγώ δεν θεωρώ πως δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα από τις συζητήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία. Δεν υπάρχουν πλέον ζητήματα τα οποία αποτελούν ταμπού ε, πριν από κάποιο καιρό η αντιπροσωπεία της ε, Ρωσίας, οι αντιπροσωπείες της αποχωρούσαν από την αίθουσα όταν θίγαμε συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό δεν συμβαίνει πια. Σε ό,τι φορά την ρωσική αντιπροσωπεία ε, αναγνωρίζουν τώρα πλέον ε, το γεγονός ότι είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται ζητήματα μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ατζέντα των συζητήσεων μας. Αλλά προφανώς και είναι δύσκολο το να αποφασίσουμε ή να πούμε ποια ήταν τα σαφή συγκεκριμένα αποτελέσματα στα οποία μας οδήγησαν αυτές οι διαβουλεύσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Νόρντλαντερ για αυτή την παρέμβαση. Ίσως θα μπορούσα να τονίσω Ε, με βάση και την η ε, ενόψη και τις διαστήσεις του ΕΣΕ σε ό,τι αφορά αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βαρσοβία, ενδεχομένως να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι από όλοι αυτή τη συζήτηση. Ε, δηλαδή θα μας δώσει κάτι τέτοιο περισσότερες ε, δυνατότητες να συνεργαστούμε με άλλα κράτη ώστε να καταπολεμήσουμε την κλωνοκρατία και ούτω καθεξής. Ε, ο κύριος Τίμαντς τώρα έχει το λόγο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας πει τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα είμαι σχετικά σύντομος αλλά θεωρώ πως η βασική ερώτηση η οποία τέθηκε από πολλούς είναι μια ερώτηση την οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε εύκολα. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Διάλογος ή άσκηση πολιτικών πιέσεων. Θεωρώ πως θα πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο, τον πολιτικό διάλογο με τη ρωσική πλευρά σε όλα τα επίπεδα. Ε, την ε, τελευταία εβδομάδα, και αν παρακολουθείτε το Σουηδική Προεδρία, αν κάνω λάθος, έγινε μια ε, συζήτηση από την πλευρά τη δικιά μα με τον κύριο Λάλμπροφ και τέθηκαν κάποια τέτοια ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ταυτόχρονα εμείς στο πλαίσιο του διαλόγου δείχνουμε μια ολόκληρη γκάμα από ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το κάναμε και στις 6 Νοεμβρίου. Από την άλλη πλευρά αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να στήσει κανεί πίεση στη Ρωσία. Και λαμβάνει κανεί την εντύπωση ότι μερικέ φορέ η άσκηση πιέσεων στη Ρωσία δημοσίω ε, μπορεί να είναι αντιπαραγωγική. Άρα λοιπόν, η δική μας προσέγγιση, δηλαδή κάνοντας δηλώσεις, ε, ε, θίγοντας αυτά τα ζητήματα σε πολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί την πιο αποτελεσματική οδό αλλά θα πρέπει να συνοδευτεί αυτός ο διάλογος από συγκεκριμένη λήψη μέτρων ε, και αυτό το συνδέω και με την εξέταση που κάνουμε αυτή την περίοδο προς το τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να βοηθήσουμε με συγκεκριμένα μέτρα τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και θα προσπαθήσουμε να βρούμε εδώ κάτι από κοινού με τις ρωσικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την ε, τρέχουσα ε, υπόθεση, δηλαδή ο κύριος ε, κατά τον κύριο Όλου ε, για να τονίσουμε ακριβώς το πολιτικό μας ενδιαφέρον και τη σημασία που δίνουμε σε αυτήν την υπόθεση. όμως θα πρέπει κανείς να πει πως δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και ορισμένες θετικές πτυχές. Αντιλαμβανόμαστε από τις ρωσικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις η σχετική νομοθεσία για αυτές οδήγησε σε κάποιες βελτιώσεις. Για παράδειγμα στο ότι μπορούν δηλαδή να εργαστούν χωρίς να τους ασκούνται τόσο πολλές πιέσεις. Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών δημιούργησε μία ειδική μονάδα για την καταπολέμηση ε, φαινομένων ρατσισμού και ναζισμού και εκεί είδαμε κάποιες επιτυχίες. Ε, πολύ πρόσφατα, αρχές Σεπτεμβρίου δηλαδή, διαπιστώσαμε ε, την ε, δημιουργία ενός ε, προγράμματος μάστερ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνεργασία και με, την, με το αντίστοιχο πανεπιστημιακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια τέτοια επιμέρους στοιχεία και θα πρέπει να συνεχίσουμε και με τις δύο όντως δηλαδή να συνεχίσουμε να στιγουσκούμε πιέσεις αλλά να συνεχίσουμε και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την κατάσταση σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τιμάντς. Ναι, τέτοιου είδους ε, μηχανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν από κοινού. Έχουμε λοιπόν ακούσει πολλές ε, πρακτικές ε, προτάσεις ως προς το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει τα δικά της ζητήματα, για παράδειγμα πώς μπορεί να ενδυναμώσει ε, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Επίσης, ε, τύχηκαν και κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις θεωρήσεις και ούτω καθεξής. Έχουμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμέ, οι οποίες ισχύουν για τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές και η τήρησή τους θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούνται στη Ρωσία, γιατί βέβαια ισχύει το γεγονό ότι πολλοί από αυτού του κανόνε, από αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ δεν πληρούνται. Δεν τηρούνται. Ε, και στο πλαίσιο αυτή τη νέα εταιρική σχέση που σχεδιάζουμε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπεριλάβουμε και ανθρωπιστικέ ρήτρε. Και βέβαια θα πρέπει να συνεργαστούμε εδώ και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Και βέβαια σε αυτό θα επανέλθουμε και στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής για τον Κάφκασο όταν θα έχουμε και τη συνάντηση δηλαδή με επιτραπέζοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα σα ευχαριστώ λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι, για όλη αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Κλείνουμε λοιπόν εδώ με το δημόσιο ανοιχτό τμήμα της συζήτησής μας. Και μπορούν λοιπόν ε, οι βουλευτέ και οι μέλη τη Επιτροπή μα να συνεχίσουν τη συζήτηση εδώ και κλεισμένο το θηρόν, αλλά δεν μπορούν ε, βοηθοί του να παραμένουν. Θα μιλήσουμε λοιπόν ε, για μία άτυπη ε, συζήτηση που έλαβε χώρα σε τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Θα κάνουμε λοιπόν ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και σας ε, ενημερώνω εκ νέου ότι το δημόσιο τμήμα της ε, σημερινής συνεδρίασης έληξε.